Ωραία, αρχίζουμε αργά, οπότε δεν θα περιμένουμε περισσότερο. Τι να κάνουμε βέβαια, όλοι προσπαθούμε να τελειώσουμε με τις δουλειές μας. Καλώς ορίζω εδώ τον Υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας. Για άλλη μια φορά έρχεται εδώ στην Επιτροπή μας προκειμένου στο τέλος της Προεδρίας της Λιθανικής, αν και όχι εντελώς το τέλος, γιατί αν μη τι άλλο όσον αφορά την ΕΚΟΝ υπάρχουν διάφορες σημαντικοί τριμερείς διάλογοι που λαμβάνουν χώρα και που προχωράμε. Ευτυχώς προχωράμε αρκετά. Λοιπόν, για 10 λεπτά ο Υπουργός και μετά θα περάσουμε σε ερωτήσεις από τους Ευρωβουλευτές που ελπίζω να μην είναι πολύ μεγάλες για να μπορέσουμε να έχουμε αρκετές ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα κάνω το γύρο των πολιτικών ομάδων, νοσήθηστε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Σάρων, ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτές της Επιτροπής αυτής. Χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι για μένα είναι δύσκολο σε 10 λεπτά να σας τα πω όλα. Ειλικρινά λοιπόν, αν κοιτάξουμε λίγο πίσω πριν από... Ξέροντας ότι φτάνουμε στα Χριστούγεννα που να είναι, αλλά πριν τα Χριστούγεννα έχουμε ακόμα μερικές μέρες εντατικής δουλειάς, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο σε διάφορους φακέλους, σε διάφορα θέματα. Όπως και να έχει το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι εκτιμά όλος ιδιαίτερος τη συνεργασία μαζί σας, την επαγγελματική, την αποτελεσματική, γιατί χωρίς τη δικιά σας συνεργασία δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό δεν το λέω μόνο γιατί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτες, αλλά επίσης γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και έτσι να δημιουργούμε κάτι από κοινού. Η Λιθωνική Προεδρία λοιπόν νομίζω ότι κατάφερε να προχωρήσει σε διάφορους φακέλους. Έξι μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Βέβαια δεν αρχίσαμε από το μηδέν, αρχίσαμε όμως με μια γερή, καλή βάση που είχαν φτιάξει προκάτοχή μας, η λαδική Προεδρία δηλαδή. Και έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε και να αφήσουμε γερά θεμέλια για την επόμενη Προεδρία, την ελληνική που αναλαμβάνει μετά από μας. Όμως θα σταθώ λίγο στα τέσσερα θέματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα της Προεδρίας μας και που σας είχα παρουσιάσει στην αρχή της Προεδρίας μας, τον Ιούλιο δηλαδή που μας πέρασε. Το πρώτο θέμα είναι η νομοθεσία για τα οικονομικά ζητήματα. Η Τραπεζική Ένωση ήταν πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη. Προτεραιότητα. that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that, uh, with that job. Uh, of... Το πιο σημαντικό θέμα που έπρεπε να αναλάβουμε υπήρχαν διάφοροι φάκελοι και χαίρομαι που την καταλήξαμε στον τριμερή διάλογο όσον αφορά την ε, τραπεζική ανάκαμψη και εξυγίανση. πολύ βασικό για ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση. Ελπίζω ότι και το Συμβούλιο πολύ σύντομα θα μπορέσει να επιβεβαιώσει την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τους τριμερείς διαλόγους. Είναι πολύ βασικό αν θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές. Όχι μόνο όμως και στους Ευρωπαίους πολίτες γιατί η δέσμευση που έχουμε αναλάβει είναι ο τραπεζικό τομέας να είναι πιο δυνατός και να προστατεύονται τα χρήματα των ε, αποταμιευτών. Είναι προτεραιότητά μας λοιπόν όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση αυτό το θέμα. Η αρχή ποια είναι. Είναι ότι όσοι εποφελήθηκαν από την ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες πρέπει να αναλάβουν και το κόστος αν τα πράγματα πάνε άσχημα. Αυτή είναι η αρχή την οποία εμείς εφαρμόσαμε στην ε, οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών. Και βάσει αυτού συνεχίζουμε και στις συνεδριάσεις του ΕΚΟΦΗΝ. Νομίζω ότι το SRM είναι ο βασικός φάκελος πάνω στον οποίο πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν είναι βέβαια κάτι τυποποιημένο, γι' αυτό ίσως μπορείτε να διαβάσετε πολλά και διαφορετικά πράγματα στον τύπο που μερικές φορές δείχνουν περίεργα ότι ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά στην νομοθεσία. Όμως νομίζω ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από το οποίο όλοι μπορούμε να εποφεληθούμε και είναι κάτι το οποίο δικαιολογεί και την δημιουργικότητα που χρησιμοποίησαμε για αυτή την υπόθεση. Είμαι αισιόδοξο λοιπόν για τις αυριανές συζητήσεις, έχοντας μάλιστα υπόψη και τις συζητήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν πολύ παραγωγικές, θα έλεγα ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Ήταν ένα σημείο καμπής μερικές φορές υπάρχει πόλωση στις χώρες μέλη. Εδώ όμως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα και έτσι η επερχόμενη ελληνική προεδρία θα αναγκαστεί να ολοκληρώσει τους τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε πριν ολοκληρωθεί ο πολιτικός κύκλος να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα. Ελίζα, εσείς θα έχετε δύσκολη δουλειά, πιστεύω. Όμως, θα μπορέσουμε και εμείς να σας βοηθήσουμε, γιατί και εμείς συμμετέχουμε στο τρίο αυτό των τριών προεδριών της ελλαδικής, της Λιθανικής και της Ελληνικής δηλαδή. Ο φάκελος αυτός νομίζω, για μένα προσωπικά, ότι είναι ο πιο σημαντικός. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Ένα άλλο πυλώνα της, Ευρωπαϊκής της ε, Ένωσης της Οικονομικής είναι το DGS. Νομίζω ότι εδώ μας μένει ένας τριμερής διάλογος. Είμαστε σε θέση να πετύχουμε συμφωνία υπό τη Λιθουανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγγύηση καταθέσεων ένα άλλο θέμα είναι η ασφάλεια των τίτλων. Είναι το MIFID, η οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Εδώ χρειάζομαι την δικιά σας στήριξη για να ολοκληρωθούν και αυτοί οι φάκελοι. Όπως κάναμε και με το Omnibus 2, την οδηγία αυτή, και με τον Μπούρχαρτ που είναι. Α, εκεί, Μπούρχαρτ. Νομίζω ότι μαζί είχαμε μεγάλη επιτυχία με το Omnibus 2. Πιέσαμε για να περάσει αυτό το θέμα, να προχωρήσει. Πράγμα που θεωρώ μεγάλο επίτευγμα, γιατί από 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο της οδηγίας Solvency 2, που αποτελεί μέρος του Omnibus 2, θα αρχίσει να ισχύει. Γι' αυτό και η οδηγία η BRD συμφωνήθηκε να προχωρήσει περισσότερο και να ισχύσει επίσης από 1η Ιανουαρίου του 2016 οδηγία δηλαδή για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών. Άρα η ημερομηνία αυτή είναι συμβολική πια. Γιατί πολύ σημαντικά θέματα μπαίνουν στο αυλάκι και αρχίζουν να ισχύουν. Είναι σημαντικό επίσης το θέμα της οδηγίας για τις υποθήκες. Ευχαριστώ που το ψηφίσατε στην Ολομέλεια. Έτσι, ολοκληρώνεται το έργο προηγούμενων οδηγιών, αλλά εμείς το ολοκληρώσαμε, εμείς βάλαμε την τελεία. Πολύ σημαντικό μήνυμα για τους πολίτες, αλλά και για τις επιχειρήσεις μας. Ναι, για τις επιχειρήσεις ΒΕΝ είναι και αυτός πολύ σημαντικός φάκελος και εδώ πιέζουμε όσο μπορούμε περισσότερο για πρόοδο. Δεν μπορώ βέβαια να υποσχεθώ ότι πριν τα Χριστούγεννα θα τα έχουμε καταφέρει, αλλά θα το προσπαθήσουμε και θα δούμε. Η οδηγία τώρα για τις πληρωμές. Και εδώ είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Την Παρασκευή, ελπίζω προχωρήσουμε επίσης όσον αφορά την νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος. Εδώ θα έλεγα ότι δεν προχωρήσαμε αρκετά, παρόλο που κάναμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Θα δούμε μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής σας, τον Ιανουάριο νομίζω του 2014, θα δούμε που θα βρισκόμαστε. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο τμήμα του πακέτου μας, που είναι θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Εδώ το ευρωπαϊκό εξάμεινο ήταν μία από τις προτεραιότητές μας. Το ΕΚΟΦΗΝ εξέτασε διάφορες πρωτοβουλίες, διάφορα ζητήματα εδώ. Για παράδειγμα, τα σχέδια, τα δημοσιονομικά που υποβάλλουν οι χώρες της Ευρωζώνης. Υποβάλλουν τα σχέδια αυτά του προπολογισμού, εγκρίνονται Βλέπουμε που υπάρχει θέμα λίματος. Υπάρχει βέβαια και η έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική ανάπτυξη. Νομίζω ότι το επόμενο εξάμεινο θα είναι κάπως ε, διαφορετικό από ό,τι είχαμε ως τώρα. Και όχι μόνο εξαιτίας της Λιθουανικής Προεδρίας, για αυτά που έκανε δηλαδή η Προεδρία μας, αλλά και χάρη στις προσπάθειες που έκαναν πολλοί παράγοντες ώστε να γίνει κατανοητό ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο βοηθάει ώστε η οικονομική διακυβέρνηση να λειτουργήσει καλύτερα και να έχει σαν αποτέλεσμα η ΟΝΕ να λειτουργεί καλύτερα. Τώρα στο θέμα της φορολογίας και εδώ επετέχθη πρόοδος. Δυστυχώς η οδηγία για τις αποταμιεύσεις η ανανομένη πρόταση δηλαδή, απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και το Κοινοβούλιο μόνο γνωμοδοτεί. Δεν πετύχαμε την ομοφωνία. Υπάρχουν δύο χώρες οι οποίες ακόμα αντιτίθενται παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. Όμως το θέμα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών εδώ αν μη τι άλλο, στο μυαλό μας προχώρησε το θέμα. Δηλαδή όλοι καταλάβαμε ότι οι προδιαγραφές ΟΣΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί και να εφαρμόσουμε πια την αυτόματη αυτή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορολογικών αρχών. Τέταρτο τμήμα. Εδώ επιτρέψτε μου να το αναφέρω, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα της δικιάς σας Επιτροπής, παρόλα αυτά Μπορώ να εκφράσω εδώ την ικανοποίησή μου που καταφέραμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουμε το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πετύχαμε να εγκρίνουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014, το συμπληρωματικό επίση για το 2013 και, και δεν πρόκειται μόνο για τα 325 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να επενδυθούν από 1η Ιανουαρίου του 2014, πρόκειται και για νέες πρωτοβουλίες. Νέες πρωτοβουλίες στον κανονισμό για την ε, πολιτική συνοχή, μεταξύ άλλων, πώς να συντεριάξουμε τα Ευρωπαϊκά Διαφορετικά Ταμεία, ε, άλλα οικονομικά μέσα, ιδιωτικές πηγές πόρων, ώστε να ενισχύσουμε την απόδοση κάθε ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που πηγαίνει στα κράτη-μέλη και πώς να υπάρξει μόχλευση 5 με 8 φορές. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που συζητήθηκαν πολύ προσεκτικά κατά το άτυπο Συμβούλιο Εκοφήν του Σεπτεμβρίου που Σάρων Πόλς ήταν παρούσα και βοήθησε πολύ με την παρουσία της εκεί ως προσκεκλημένη επίσημη. Και συνεχίζω στα λιθουανικά, λέει ο Υπουργός. Βάλτε τα ακουστικά σας. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας, που ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική, πολύ χρήσιμη, αλλά και πολύ ευχάριστη. Είμαι πεπισμένος ότι οι προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας, δηλαδή μια ανοιχτή Ευρώπη, αξιόπιστη, σε ανάπτυξη, αυτές οι προτεραιότητες πιστεύω ότι επιτεύχθηκαν. Και επιτεύχθηκαν χάρη στις αποφάσεις που πήραμε από κοινού. Είναι πιο βιώσιμη πια η Ευρώπη. Βλέπουμε ότι η οικονομία ξεκινάει με νέο βήμα και η Ευρώπη είναι πια πιο ανοιχτή. Η Προεδρία μας πιστεύω ότι αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση πρώτα απ' όλα για τη Λιθουανία, για τη χώρα μου, γιατί μας δόθηκε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Μπορέσαμε έτσι να διαπιστώσουμε κι εμείς ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε πολλά πράγματα και ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά εφόσον δρούμε από κοινού. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμικό όργανο και ευχαριστώ πολύ όλους ιδιαίτερους στη δικιά σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, μετρούσα πόσους φακέλους είπατε ότι θα κλείσετε. Αν όλα πάνε καλά αυτή τη βδομάδα, κάπου 10 φακέλους της Επιτροπής μας θα κλείσετε οικονομικούς. Καλό ρεκόρ αυτό. Δεν ξέρω κατά πώς θα τα καταφέρετε βέβαια, αλλά όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, σίγουρα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι τεράστια όπως είπατε κι εσείς, για πολλές και δύσκολες μάλιστα υποθέσεις και ορισμένες αποθέσεις είχαν κολλήσει για πολύ καιρό. Λοιπόν, τώρα περνάμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. ΕΛΚ πρώτα απ' όλα, ο Ζαν Πολ Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Νομίζω πραγματικά ότι πρέπει να σας συγχαρούμε. Και όντως σας συγχαίρουμε, η μεν και η δε, γιατί ο απολογισμός της Προεδρίας σας είναι εξαιρετικός, το είπε και Αν όλα πάνε καλά, όντως θα έχουμε κλείσει δέκα νομοθετήματα, δέκα σημαντικά θέματα Φαντάζομαι ότι όταν αναλάβατε τις αρμοδιότητές σας δεν φανταζόσασταν ούτε κι εσείς ότι θα καταφέρατε να πετύχετε τέτοιο σημαντικό αποτέλεσμα. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε στο δικό μου το γραφείο ήσασταν και αισιόδοξο, αλλά είχατε και μια κάποια ανησυχία. Εγώ σα είχα πει τότε ότι ήμουν απεπισμένο ότι η δική σα προεδρία θα ήταν πολύ καλή και όντω το αποδεικνύει τώρα και η πραγματικότητα. Συγχαρητήρια λοιπόν για την εξαιρετική δουλειά που έχετε επιτελέσει σε μια δύσκολη περίοδο για ζητήματα πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι η Προεδρία σα η Λιθουανική επέτρεψε στην Ευρώπη πραγματικά να σημειώσει πρόοδο και καταφέρατε τελικά να αποκρισταλώσετε σε όλε τι συζητήσει που είχαμε όλε αυτέ τι θετικέ ενέργειε για διάφορα ζητήματα όπω το ζήτημα με το οποίο ασχολείται ο κύριο Μπούρχαρτ, ο οποίο συνεργάστηκε πολύ μαζί σα. Δεν έχω να σα υποβάλω αυτή τη στιγμή κάποια σημαντικά ερωτήματα. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στην Τραπεζική Ένωση που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα μπορούσατε κι εσείς μιλώντας την δική σας τη γλώσσα να μας πείτε πώς πιστεύετε από προσωπικής πλευράς ότι μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε μια κατάλληλη λύση σύντομα για το ζήτημα της Τραπεζικής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα κάνατε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Uh, <laughs> <laughs> ε, ε, ε, ε, ε, thank Σας ευχαριστώ, Ζαν Πολ, για τις πολύ καλές αυτές ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο με δικά μου λόγια και στη δική μου γλώσσα να σας πω εγώ ακριβώς ε, τι πρέπει να γίνει, ποιους συμβιβασμούς θα πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε. Και πρέπει να σας πω απολύτως ειλικρινά ότι προσπάθησα εγώ να πετύχω τέτοιους συμβιβασμού ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Γίνανε πάρα, πάρα πολλές συζητήσεις, διμερείς, πολυμερείς, διαβουλεύσεις. Είχαμε διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις. Πολλές φορές πρέπει να σας το πω ότι είχαμε και πραγματικές συγκρούσεις, όχι κινηματογραφικές αναγκαστικά, αλλά όντως διεξήχθησαν πολύ δύσκολες συζητήσεις ορισμένες περιστάσεις. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε υποβάλει κάποιες προτάσεις οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή μπορούν να επιφέρουν κάποιες αλλαγές ή πολλές φορές τροποποιούνται και οι ίδιες οι προτάσεις μέσα σε κάποιες ώρες, όχι μόνο από τη μία μέρα στην άλλη. Ζαμπό, λοιπόν, δεν θα ήθελα να επισέλθω αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα και δεν έχουμε συμφωνήσει επ' όλων των λεπτομεριών. Έχουμε πει μεταξύ μόντων των Υπουργών ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα μέχρι να αποφασιστούν όλα. Αυτή είναι η βασική μας αρχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω πάντως ότι αύριο θα είμαστε σε θέση να τοποθετήσουμε τα πάντα στη σωστή τους θέση. Θα έχουμε πολλά διαφορετικά έγγραφα, θα σας κοινοποιήσουμε τα πάντα. Ενδεχομένως να μην μπορούμε να διαπραγματευτούμε επόλων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα τα ζητήματα. Θεωρώ πάντως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να δει και να αξιολογήσει οτιδήποτε έχει αποφασιστεί ή πρόκειται να αποφασιστεί στο μέλλον. Λυπάμαι που είμαι ασαφή στην απάντησή μου. Θα δώσουμε το λόγο στην Ελίζα σε λίγο. Αν όντω αλλάζουν τα πράγματα κάθε δύο ώρε, τότε α αλλάξουν προ την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν μη τι άλλο. Πιστεύω ότι θα ήταν πραγματικά δυστυχές, ατυχές αυτή τη στιγμή και μια τεράστια καταστροφή αν τελικά κινηθείτε προς μια κατεύθυνση που δεν θα ήταν τόσο δημοκρατική και που θα άφηνε εκτός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμένω στο σημείο αυτό και νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα ατυχές το τέλος της Προεδρίας σας αν καταλήγαμε σε κάτι τέτοιο. Παράκαμψη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελίσσα, Σε ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή που έκανες ε, Σάρον. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και την Προεδρία. Θεωρώ πραγματικά ότι έχετε επιτελέσει ένα πολύ καλό έργο. Με τη δική σας άλλωστε την Προεδρία αρχίσαμε να συζητάμε την λειτουργία της οικονομικής διακυβέρνησης καθώς επίσης και τις επιμέρους λεπτομέρειες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέρατε να καταλήξετε σε μια συμφωνία όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία και όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές. Βέβαια, λυπάμαι και εγώ που στα πλαίσια της νομοθεσίας για τα διαρθρωτικά ταμεία έχουμε την μακροοικονομική αιρεσιμότητα που θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι που αντιβαίνει στην ίδια την νομοθεσία. Έχετε κάποιες βασικές αρχές ισότητας και δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι πολύ καλή όσον αφορά τώρα τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία με αφορούν εμένα περισσότερο. Θεωρώ ότι η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών ήταν μια πολύ πολύπλοκη οδηγία και όντω αναγνωρίζω την πολύ σημαντική εργασία η οποία έγινε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και όλη την ομάδα διαπραγματεύση. Θα ήθελα βέβαια να μπορούσα να έλεγα τα ίδια θετικά πράγματα και για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Γιατί πρόκειται πραγματικά για ένα από τα πιο πολύπλοκα ζητήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε και θα κρυθούμε για τον ενίο μηχανισμό εξυγίανσης, για τον τρόπο που θα τον θεσπίσουμε. Όχι μόνο ο φάκελος αυτός είναι θεμελιώδης, αλλά είναι και μια πραγματική καινοτομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να στήσουμε σωστά το νέο αυτό σύστημα. Δεν ξέρω λοιπόν αν όντως τα πράγματα παρουσιάζουν μια τέτοια εξέλιξη, αν είναι τόσο ευμετάβλητα, όπως είπατε κάθε δύο ώρες. Ελπίζω, όπως το είπατε και εσείς, να προσπαθείτε όντως να πετύχετε μια καλή συμφωνία και ένα καλό συμβασμό. Ακούμε όμως τώρα κάποιες φήμες που λένε ότι ενδεχομένω η θέση του Συμβουλίου να τροποποιηθεί. Λένε ότι ενδεχομένως η τελική τοποθέτηση του Συμβουλίου να αντιβαίνει εντελώς τις βασικές αρχές που θέλουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προασπίσουμε. Ξέρετε ότι εμείς θα ψηφίσουμε σήμερα την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι αυτό θα εμπνεύσει αν μη τι άλλο και το Συμβούλιο να καταλήξει τελικά σε μια τοποθέτηση η οποία θα είναι θετική όσον αφορά το πλαίσιο που θα πρέπει να δημιουργηθεί για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Επί του παρόντος εμείς θέλουμε να σπάσουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στις τράπεζες και το δημόσιο χρέος και κατά αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να προστατεύσουμε περισσότερο τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Να μην χρειαστεί δηλαδή αυτός να πληρώνει το τίμα στο μέλλον κάθε φορά που χρεοκοπεί μια τράπεζα. Ανταυτού θα πρέπει να έχουμε ένα ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτεί πλέον τις τράπεζες οι οποίες είναι βιώσιμες αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς θα χρηματοδοτείται και το ταμείο αυτό, τι πιστώσεις θα έχει το ταμείο αυτό. Οι εισφορές θα πρέπει να γίνουν από τον ίδιο τον παραγωγικό κλάδο θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο και μοναδικό σύστημα. Μιλάμε για ενιαία εποπτεία, ενιαία εξυγίανση και για ένα ενιαίο λοιπόν ταμείο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε να αποφύγουμε με κάθε δυνατό τρόπο οποιαδήποτε πολιτική δέσμευση και καθοδήγηση όσον αφορά τη χρεοκοπία μιας τράπεζας. Αυτές είναι οι βασικές ανησυχίες λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ακούγονται αυτή τη στιγμή κάποιες φήμες που λένε ότι ενδεχομένως το ταμείο αυτό να βασίζεται σε μια διακυβερνητική συμφωνία και όχι στην κοινοτική μέθοδο που θέλουμε εμεί λέγεται ότι μπορεί να προκύψουν τελικά κάποιες ε, διακυβερνητικές ε, διατάξεις οι οποίες θα επικρατήσουν τη κοινοτική μεθόδου και αυτό μας προκαλεί μια πολύ σημαντική ανησυχία. Ελπίζω λοιπόν ότι η φανταστική αυτή ε, εργασία που έχετε επιτελέσει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας δεν θα υπονομευτεί τις τελευταίες αυτές ημέρες της Προεδρίας σας για το φάκελο αυτό. Σας καλούμε λοιπόν πολύ στεναρά να διαπραγματευτείτε ένα πολύ καλό συμβιβασμό και για αυτό το θέμα, όπως το κάνατε για πολλά άλλα θέματα. Καταλαβαίνω το ζήτημα αυτό είναι τόσο σημαντικό που πραγματικά δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αποτύχει στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Ελίζα, ευχαριστώ. Ξεκίνησες με κάτι που ίσως στην δική μου εισαγωγή δεν ανέφερα. Φυσικά Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην ομάδα μου, ιδιαίτερα ευγνώμων σε αυτούς επίσης. Ήταν μια ομάδα ιδιαίτερα πεπειραμένων και αφοσιωμένων ανθρώπων. Οι πιο έμπειροι και αφοσιωμένοι που θα μπορούσα να είχα ευχηθεί ποτέ. Πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσω, να τους ευχαριστήσω. Αλλά ας μην παραμείνουμε σε φήμες και ψιθύρους. Αλλά ασχοληθούμε με τις αρχές που απαριθμίσατε και προσυπογράφω κάθε μια από αυτές τις αρχές που απαριθμίσατε. Η διασύνδεση μεταξύ χρέους και τραπεζών θα πρέπει να πάψει να υφίσταται και αυτό είναι το κυριότερο θέμα όταν θέλουμε τώρα να δημιουργήσουμε την Τραπεζική Ένωση. Το να ξεπεράσουμε τον τομεακό κατακαιρματισμό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πραγματικά ανάγκη, αναγκαιότητα. Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης είναι ένα από τα βήματα. Ίσως όχι ένα άμεσο βήμα που θα ακολουθήσει αμέσως η άρση των ε, διαφορετικών αυτών ορίων σε σχέση με τα κράτη-μέλη, αλλά μια σταδιακή βήμα προς βήμα προσέγγιση θα πρέπει να δούμε αν θα είναι παραγωγική και πώς. Για να μπορούσαμε να πετύχουμε μια συμφωνία, να ισχύσει το bail-in, η διάσωση εκ των ένδων, εκ των έσω, ώστε να μπορέσουμε από το 2016 να προχωρήσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο απέρευσε ακριβώς από τις συζητήσεις και τους τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπέρασμα. Τώρα, στη συνέχεια, τα χρήματα, τα κονδύλια ή τα μέτρα για την επίλυση τραπεζικών προβλημάτων το πώς θα χρηματοδοτηθούν από πλευράς μας ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη και υπόσχομαι ότι θα παραμείνουμε σε αυτή την ιδέα για αυτό, την επίλυση αυτού του προβλήματος. Μια πολύ σημαντική ιδέα είναι ότι πολιτικές και άλλες εθνικές θα έλεγα ε, αρχές ή παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να επιληθεί το πρόβλημα. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε την αρχή με συνέπεια και συνεκτικότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν την Τραπεζική Ένωση. Αλλά και πάλι δεν θα ήθελα να υπησέθω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Okay, Εντάξει. Και τώρα για την Άλντε, Wolfgang, έχετε τον λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου στα συγχαρητήρια των συναδέλφων προς εμάς. Γνώρισα διάφορα μέλη των ομάδων σας και πρέπει να ομολογήσω έχουμε ένα εξαιρετικό συνδυασμό μεταξύ τεχνικής εμπειρίας και πείρας και προσωπικής αφοσίωσης και αυτό πρέπει να τύχει ρητή αναφορά και αναγνώριση. Τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω ήδη διατυπώθηκαν. Θα διατυπώσω άλλα ερωτήματα. Πρώτον, πιστεύετε ότι οι προποθέσει για μη μέλη τη Ευρωζώνη να συμμετάσχουν εθελοντικά στην Τραπεζική Ένωση έχουν καλά επιλεγεί. Υπάρχουν αυτέ οι προποθέσει και είναι δεδομένε ή βλέπετε κάποιο κίνδυνο να διαγράφεται Ότι de facto η Ευρωζώνη ναι μεν θα ολοκληρωθεί περισσότερο αλλά θα υπάρξει ένας διχασμός μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, και των υπόλοιπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχουν σε αυτή. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, αναφέρθηκε ήδη αυτή η θα έλεγα επιζήμια εξάρτηση τραπεζών, τραπεζικών θεμάτων και κρατικών ομολόγων και κρατικού χρέους. Θέλουμε αυτό να το διαχωρίσουμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα βλέπουμε ότι διαθέτει κονδύλια με πολύ χαμηλά επιτόκια και χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα από τις τράπεζες στα κράτη-μέλη για να επενδύσουν σε κρατικά ομόλογα. Δηλαδή επιτυγχάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Και τώρα μέσω της ε, quality review ε, όπου αυτά τα κρατικά ομόλογα ίσως με περισσότερο κριτικό φως ε, και κριτικές παρατηρήσεις αντιμετωπίζονται ίσως αυτό μπορεί έτσι να επιληθεί σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Okay. Of course. Μάλιστα. Εντάξει. Φυσικά μία από τις αρχές της Τραπεζικής Ένωσης όπως και στο SSM που και αυτό με επιτυχία ολοκληρώσαμε δεν ήταν απόλυτα δικό μας αυτό το χαρτοφυλάκιο πλήρως, αλλά ήταν τιμή μου να εγκριθεί αυτό τον Οκτώβριο στο ΕΚΟΦΗΝ τότε υπό τη δική μας Προεδρία και για την αμοιβαία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πάλι επίσης εδώ το Ευρωκοινοβούλιο Κοινοβούλιο μη είχε και ανταλλαγή ε, απόψεων και πληροφοριών. Όπως ξέρετε οι μη χώρες Ευρωζώνης μπορούν να έχουν ε, opt-in, εθελοντική συμμετοχή στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Και για το δεύτερο πυλόν ακριβώς ε, της Τραπεζικής Ένωσης σε αυτό το θέμα πρέπει να αντανακλά την δομή της εποπτείας και επιτήρησης με σωστό τρόπο. Πρέπει το ένα να ταιριάζει στο άλλο. Και για τις προτάσεις SRM άμεσες αναφορές ε, στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό υπάρχουν και για τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Μπορώ να σας διασφαλίσω λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών θεωρούν ότι όχι μόνο η Τραπεζική Ένωση δεν είναι μόνο προϊόν για τις ε, χώρες Ευρωζώνης Φυσικά υπάρχουν οι φυσικές πρώτες βάσεις ως ή θεμέλια πως θα ξεκινήσουμε με αυτές τις χώρες της Ευρωζώνης. Αλλά μετέπειτα στην επόμενη φάση θα υπάρξει επέκταση, διεύρυνση και σίγουρα πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για τις χώρες μη Ευρωζώνης, εκτός Ευρωζώνης που επιθυμούν να ενταχθούν στην Τραπεζική Ένωση να το κάνουν. Αλλά είναι και ένα ισοδίκαιο πεδίο δράσης ε, και δραστηριοποίησης εντός Τραπεζικής Ένωσης και εκτός Τραπεζικής Ένωσης πανενωσιακά. Αυτό το ισοδίκαιο πεδίο δραστηριοποίηση πρέπει να διασφαλιστεί και να θεμελιωθεί. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτέ τι αρχέ. Δεν είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό, διότι υπάρχει συντριπτική επιβολή της Πριτανία της άποψης ότι θα έλεγα συνένεση συνολική από όλα τα κράτη-μέλη επ' Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιτόκια, πολιτική καθορισμού επιτοκίων. Δεν έχω δικαίωμα να το κάνω αυτό και δεν θεωρώ ότι ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ έχω κάποιες αρμοδιότητες αυτή τη στιγμή να, κάνω, να πράξω κάτι τέτοιο. Όμως για την quality review, την ε, ε, αναθεώρηση για την ποιότητα, αξιολόγηση ποιότητας είναι η πρώτη φάση για την εφαρμογή του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Και αυτή η asset review θα διεξαχθεί κατά το επόμενο έτος 2014. Μέχρι ότου να αρχίσει να ισχύει πλήρως ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός την 4η Νοεμβρίου 2014. Και έτσι τα κράτη-μέλη αλλά επίσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίσης όμως και ε, εποπτικές αρχές και σώματα στα κράτη-μέλη προετοιμάζονται με ιδιαίτερη προσοχή για όλα αυτά. Η Asset Quality Review δεν είναι το μόνο εγχείρημα που έχουμε. Έχουμε και δοκιμασίες ε, ε, stress tests που θα διεξαχθούν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, European Banking Authority. Δεν υπησέρχομαι σε λεπτομέρειες. Θέλω μόνο να σας πω ότι τα μαθήματα τα οποία συναγάγαμε και μάθαμε το 2011 σε σχέση με τα tests, stress tests που έγιναν τότε, με τις δοκιμασίες τραπεζικές και άλλες που έγιναν τότε, μάθαμε ότι αυτό το εγχείρημα θα είναι πιο επιτυχές, θα στέφεται με μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά και την σωστή επικοινωνία που πρέπει να επιτευχθεί. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως γνωρίζετε, η επικοινωνία είναι σημαντικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό πώς περνάτε το μήνυμα, πώς μιλάτε για τα χρήματα, για τα κονδύλια και τις διαργασίες, για τη σωστή λειτουργία των χρηματοοικονομικών και πιστοτικών ιδρυμάτων. Okay, uh, uh, Εκ μέρους των Πρασίνων, ο Σβέν τώρα. Εσένα έχω στον καταλογό μου ως επόμενο. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εκεί, αν πάση περιπτώσει, λέει ο κύριο Γκυγόλτ. Θα ήθελα να πω μπράβο για όσα καταφέρατε. Η προεδρία σα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Εδώ βέβαια δεν είμαστε για να μετρήσουμε τα αποτελέσματα σε κάθε φάκελο χωριστά. Καταφέρατε να προχωρήσετε πολύ Και πολλοί συνάδελφοι νομίζω ότι έχουν πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα συνεχίσει η πρόοδος αυτή και τους επόμενους μήνες. Πέραν αυτού όμως. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις οικονομικές υπηρεσίες, όπου έχουμε τις διαδικασίες συναπόφασης και τους άλλους τομείς. Το αναφέρεται και ίδιος. Φορολογία, για παράδειγμα. Αν συγκρίνω το αποτέλεσμα του Μαΐου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με η ισχυρή δέσμευση να προχωρήσουμε και την έκθεση του ΕΚΟΦΗΝ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας, όπου το ΕΚΟΦΗΝ προσπαθεί κάπως έτσι σαφώς να πει ότι λίγη πρόοδος επιτεύχθηκε. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την φορολογία καταθέσεων, πρόκειται και για την φόρο αποφυγή μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων για κάθε χώρα τον Μάιο εσείς αναλάβατε δέσμευση, τώρα όμως αυτό έχει καταστραφεί μετά από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στο Συμβούλιο αν μη τι άλλο. Εδώ βλέπω μεγάλο κίνδυνο. Εδώ το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο περιορισμένο. Υπάρχουν και διάφορες γραπτές ερωτήσεις προς εσάς. Εμείς θέλουμε γραπτή απάντηση. Να ξέρουμε πότε θα την πάρουμε αυτή την απάντηση επιτέλους. Το ίδιο ισχύει και για το μέλλον της Ευρωζώνης. Αν δείτε τι δεσμεύσεις αναλήφθηκαν στο παρελθόν και πόσο λίγα αποτελέσματα έχουμε σήμερα, θα θυμόσαστε και τον Φαν Ρομπάι που υπέγραψε με τον Παρόσο και τον Τράγκη. Τελικά, ελάχιστα πράγματα επιτεύχθηκαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει μόνο το CCI. Πέραν αυτού όμως, ελάχιστα έχουν επιτευχθεί. Εντάξει, μπορεί να μην είναι δικιά σας η ευθύνη, γιατί είναι στο Eurogroup και εσείς στο μέλλον θα είσαστε μέλη εκεί. Αλλά αν μη τι άλλο βλέπουμε ότι όπου υπάρχει η συναπόφαση καταφέρνετε να προχωρήσετε πολύ. Ενώ εκεί που δεν έχουμε πλήρης εξουσίες συναπόφασης, το Συμβούλιο μπλοκάρει με συνένεση μεταξύ τους την οικονομική διακυβέρνηση τελικά στην Ευρωζώνη ή την φορολογία όπου και εκεί η πρόοδος είναι πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό και λέω ότι ανησυχώ πολύ για την ελάχιστη πρόοδο στο ΕΚΟΦΗΝ όσον αφορά την φορολογία. Τέλος, εσείς πώς βλέπετε τις εξελίξεις, δηλαδή για το SRM, για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εξυγίανση, κάποιες χώρες συναντιόνται στο Βερολίνο εκτός συνήθων διαδικασιών. Εσείς πώς βλέπετε ως Προεδρία αυτό το γεγονός. Ο Προεδρεύων, θα αρχίσω από την αρχή. Έχετε δίκιο ότι η πρόοδος σε θέματα φορολογίας δεν είναι τόσο εντυπωσιακή. Πολλοί είναι οι λόγοι. Βέβαια δεν συμφωνώ μαζί σας ότι δεν υπήρξε πρόοδος. Υπήρξε για την φορολογία. Έχετε δίκιο ότι χρειάζεται ομοφωνία και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Εδώ μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο εμπόδιο και αυτό είναι ο πολιτικό κύκλος της κάθε χώρα. Μεταξύ τους δεν συμπίπτουν οι πολιτικοί κύκλοι. Σε αυτό το εξάμεινο έχουμε δύο χώρες όπου τελείωσε ένας πολιτικός κύκλος και ο επόμενος πολιτικός κύκλος δεν άρχισε αμέσως μετά. Αυτός λοιπόν ίσως να είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η οδηγία για τις αποταμιεύσεις κόλλησε. Παρά τις έντονες συζητήσεις που είχαμε και τις αποφάσεις που ελήφθησαν πολλές φορές στο ΕΚΟΦΗΝ. Στον τομέα του ΦΠΑ πρέπει να σας πω ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα θέματα. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα υπάρξει συνέχεια πάνω στους φακέλους αυτούς. Μερικές φορές στον τομέα της φορολογίας τα θέματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα τεχνικά μιλώντας, άρα χρειάζεται να έχουμε ενημέρωση και για τα τεχνικά στοιχεία. Αυτό το οποίο εγώ τονίζω είναι ότι αλλάζει νοτροπία όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Πάντως τις ερωτήσεις σας τις έχουμε και θα απαντηθούν γραπτά και γι' αυτό σας διαβεβαιώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Εδώ διαφωνώ απόλυτα μαζί σας για το ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Φυσικά και θα είχαμε προτιμήσει και εμείς να έχουμε κανονισμούς ή τέλος πάντων κάποιες νομικές πράξεις για τον εξάντε συντονισμό των μεταρρυθμίσεων. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Από την άλλη, έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που είναι σχετικά καινούριο θεσμός παρόλο που είμαστε στο τέταρτο. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται εδώ και μερικού μήνε. Έχουμε την πρώτη αξιολόγηση των προπολογισμών των χωρών της Ευρωζώνης. Οι διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον επόμενο χρόνο έχουν ε, συμφωνηθεί και είναι κάπως διαφορετική από το 2013. Από τη μια επισημοποιείται περισσότερο, τυποποιείται περισσότερο, αλλά δεν είναι πιο περίπλοκο. Αυτή είναι μια άλλη ιδέα, βλέπετε, που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, ότι δηλαδή δεν θέλουμε να περιπλέκουμε τα πράγματα, αλλά να μπορούμε να έχουμε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες. στο ευρωπαϊκό δηλαδή εξάμεινο να μην γίνεται τόσο τυποποιημένο. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα για αύριο ή τα Χριστούγεννα, αλλά όταν συζητηθούν τα εθνικά ε, προγράμματα ε, σταθερότητας το... την Άνοιξη, θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν τα φετινά αποτελέσματα με τα προηγούμενα και ήδη θα δείτε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Η έκθεση αυτή πάει πολύ περισσότερο στο βάθος. Κάτι πολύ θετικό. Είναι μια προσέγγιση βήμα-βήμα. Εντάξει, μπορεί να θέλαμε, όπως είπα και νωρίτερα, να έχουμε νομικές πράξεις. Δεν έχουμε. Ιδεολογικά όμως, στο μυαλό μας, όπως είπα και πριν, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε προχωρήσει. Έρχομαι τώρα στο Eurogroup. Εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί ήμουνα ο πρώτος πρόεδρος ΕΚΟΦΗΝ στην ιστορία που προέρχομαι από μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη. Όμως συμμετείχα στις συζητήσεις για διάφορα ειδικά ζητήματα. Υπήρχαν διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη για τα οποία μου ζητήθηκε η παρουσία. Κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα το Eurogroup που προβλέπεται στη συνθήκη και το ECOFIN να συνεργάζονται πολύ πιο αποτελεσματικά. Ήταν πολύ χρήσιμο και για μένα, ομολογώ. Και προσβλέπω το Σεπτέμβριο που μας έρχεται να ξαναπάω, βέβαια με διαφορετικό νομικό καθεστώς πια. Είμαι πολύ αισιόδοξο. Πάντως όλοι οι σχηματισμοί αυτοί στο Συμβούλιο μπορούν να συνεργαστούν και μπορούν να προσφέρουν ενδιαφέρουσες ιδέες και καρποφόρες. Αυτό ισχύει και για τις συναντήσεις τις οποίες αναφερθήκατε. Δύο, τρεις ή τέσσερις ή παραπάνω υπουργοί. Είναι μια πρακτική ιδιαίτερα χρήσιμη για να ευθυγραμμίζονται οι θέσεις, γιατί όταν είμαστε και 28, ο κίνδυνος είναι να μην καταλήξουμε καθόλου σε αποτέλεσμα. Οπότε ήταν δικιά μου προσωπική θέση, ήδη από την αρχή, από τον Ιανουάριο δηλαδή φέτος, να ενθαρρύνω τις προσωπικές επαφές με όλους τους συναδέρφους. Είδαμε καλά αποτελέσματα από τέτοιες επαφές έγιναν πολλές τέτοιες επαφές και διμερείς και πολυμερείς με πολλούς συναδέρφους μου. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να προετοιμάζονται οι αποφάσεις. Βέβαια, όλοι συμφωνούμε, όλοι οι σχηματισμοί, όλοι οι διμερείς ε, και πολυμερείς επαφές που είχα, έδειξαν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο τραπέζι του ΕΚΟΦΗΝ. Οι νομικές αποφάσεις, οι νομικές πράξεις. λαμβάνονται στο ΕΚΟΦΗΝ και από άλλου. Και επιμένω σε αυτή τη θέση. Οι συνάδελφοί μου το καταλαβαίνουν επίσης πολύ καλά και συμφωνούν μαζί μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Από το ECR τώρα ο κύριος Έπινγκ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, κάποιες συγκεκριμένες λίγες ερωτήσεις πρώτα ερώτηση σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση. Ποιο αποφασίζει για την επίλυση ε, για την ε, αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος στο ESM, το SSM, η διοίκηση της ε, Κεντρικής Τράπεζας, το ΕΚΟΦΗΝ, Ποιο Δεύτερον, όσο αφορά το backstop, είσαστε υπέρ μιας τομεακής αντιμετώπισης ω θέμα θεωρία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Καταλήγω στο συμπέρασμα όμω ότι αυτό θα συμπεριλαμβάνει μόνο 55 δις ε, ευρώ μέχρι το 2025-2028 και θα είναι πολύ μικρό αυτό το ποσό και με μεγάλη καθυστέρηση και όταν μία ή δύο τράπεζες θα είναι σε μεγάλο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα θα είναι σαν πυροσβεστική χωρίς νερό να σβήσει τη φωτιά Ποια θα ήταν η δική σας ε, επιλογή, προτίμηση, δημόσιο backstop είναι ένα δίκτυο ε, ταμείων διάσωσης ή ένα ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης ή το ESM. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσαφινιστεί αυτό. Θέλουμε να προστατέψουμε τους φορολογούμενους και στο τέλος τέλος ε, θα δούμε ότι θα είναι τόσο μικρό το ε, επίπεδο διάσωσης που θα πρέπει να συμπληρωθεί με άλλες μεθόδους διάσωσης. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε τις απόψεις για το διαχωρισμό λιανικών υπηρεσιών, λιανικής τράπεζας εντός εισαγωγικών ε, σε σχέση με τον κανόνα Volcker Rule που συζητείτε. απάντηση. Έχετε πολλές συγκεκριμένες εξειδικευμένες ερωτήσεις για τις οποίες είτε δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση είτε δεν θα μπορούσα να απαντήσω και υπό ηθικής πλευράς ε, ως προεδρεύων της, ε, του ΕΚΟΦΗΝ υπό αυτή την αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε πολλές από τις ερωτήσεις, όμως αποφασίσαμε μία αρχή να ισχύει όσον αφορά το backstop για το backstopping, τον προστατευτικό μηχανισμό, για το πώς δηλαδή στις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τον τραπεζικό τομέα θα πρέπει να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Πρώτον, η πρώτη πηγή είναι πάντα ο ιδιωτικός τομέας ο οποίος θα πρέπει να υπομίζεται το βάρος ε, και τον, τις συνέπειες των αποφάσεων για την ε, αναδιάρθρωση για να βοηθηθούν τράπεζες και να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Η πρώτη πηγή λοιπόν πάντα θα είναι ο ιδιωτικός τομέας είτε σε σχέση με την ανακεφαλοποίηση είτε κάποια δυνατότητα διάθεσης ε, ε, ε, από πλευράς τους. Η δεύτερη πηγή θα είναι κρατικές, ε, θα είναι κρατική άντληση χρημάτων, δημόσια δηλαδή υποστήριξη από τα κρατημέλη. Και η τρίτη φάση, μόνο στην τρίτη φάση θα έρχεται κάποια ευρωπαϊκή πηγή άντλησης ε, ε, κεφαλαίων για να βοηθήσουν. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ποιος θα λαμβάνει την απόφαση, ποιος θα κάνει τι, ποιος θα πληρώνει τι και πώς θα συμμετέχει, είναι ακριβώς θέμα περαιτέρω συγκεκριμένων κανονισμών και διατάξεων σε σχέση με τη δική σας ερώτηση, το SRM για παράδειγμα, ίσως ε, εδώ θα ε, εντασσόταν ε, και έχουμε ήδη μια απάντηση ποιος θα επιλύει τα προβλήματα τραπεζών ή θα είναι η Εθνική Αρχή Επίλυσης Τραπεζικών Προβλημάτων και στο SRM στην Τραπεζική Ένωση ακόμα δεν έχω μια τελική καθοριστική απάντηση αλλά μετά από το συμβιβασμό που θα επιτευχθεί αυτή θα είναι μια πρόταση στο τριμερή διάλογο που θα καταλήξουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάποια ρύθμιση. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, διαχωρισμό λιανικών, υπηρεσιών ε, λιανικών, εξατομικευμένων υπηρεσιών ε, και ε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω παρά μόνο ατομικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούκαρτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και εγώ από πλευράς μου θα ήθελα ρητά να σας εκφράσω ευχαριστίες για το έργο που επιτελέσατε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Πιστεύω ότι πραγματικά εξαιρετικό έργο επιτελέσατε και εδώ παρεμβαίνω ιδιαίτερα για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε αναφέρθηκαν από εσά μετά από 13 έτη διαπραγματεύσεων μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε και το θέμα Omnibus. Σας ε, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες γι' αυτό. Τρεις ερωτήσεις θα είχα να διατυπώσω που σήμερα θα ήθελα να σας απευθύνω. Αφενός, πολλά καταφέραμε κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας. Πιθανόν βέβαια 10 χαρτοφυλάκια ολοκληρώνονται με αυτόν τον τρόπο. Ερώτησή μου, πώς βλέπετε εσείς και πώς εκτιμάτε τα επόμενα έτη ως σημαντικά νομοθετικά χαρτοφυλάκια με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Ποια θα είναι αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Η χώρα σας, εσείς ο ίδιος ως Υπουργός Οικονομικών της ε, Λιθουανίας θέλετε να προσχωρήσετε στο ευρώ πράγμα το οποίο το καλωσορίζω και το χαιρετίζω θερμά. Θα μπορούσατε να κάνετε κάποιε παρατηρήσει, κάποια σχόλια. Πώ βλέπετε αυτή τη στιγμή την κατάσταση σε σχέση με το ενιαίο νόμισμα. ποιε μεγάλε προκλήσει ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με το 2014, ε, σε σχέση με το ευρώ, την ευρωζώνη και αυτό το εγχείρημά σα. Τρίτη ερώτηση, σε σχέση με τον φόρο χρηματο, ε, χρηματικών συναλλαγών. Πώς ε, εκτιμάτε το τέλος ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, πώς βλέπετε την προοπτική εισαγωγή αυτού του τέλους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε σε αυτά τα τρία ερωτήματα να τοποθετηθείτε, θα σας ήμουν ευγνώμων αν το κάνατε. Ευχαριστώ. Well, σας... Θα ήθελα να σας πω λοιπόν όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση για τα σημαντικά χαρτοφυλάκια στον χρηματοοικονομικό τομέα. Πιστεύω ότι είχαμε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ το Σεπτέμβριο. Δεν λάβαμε αποφάσεις τότε σε αυτό το ΕΚΟΦΗΝ. Όμως υπήρχαν κάποιες οδοί, κάποιοι διάβλοι προς το μέλλον που συζητήθηκαν και εξετάστηκαν στις διαβουλεύσεις μας και που φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικές. Ένα από τα θέματα ήταν η μελλοντική αρχιτεκτονική του τομέα αυτού στην Ευρώπη στο μέλλον. Πιστεύω ότι πολλά έχουμε να πράξουμε. Παρότι υπάρχουν πολλά τεχνικού χαρακτήρα θέματα ως τα χαρτοφυλάκια που βρίσκονται επί τραπέζης, πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρωθούν και πρέπει να καταφέρουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ολοκληρώσουμε όμως η μεγαλύτερη, βαθύτερη κατανόηση για τον χρηματοοικονομικό τομέα, πώς αυτός θα πρέπει να διαμορφωθεί και να δομηθεί, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίκαιρο θέμα για την Ευρώπη. Παράδειγμα, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το θέμα το οποίο παρουσιάστηκε και από την Ιρλανδική Προεδρία συζητήθηκε τον Απρίλιο στο Δουβλίνο, στο άτυπο Εκοφίν υπό την Ιρλανδική τότε Προεδρία. Προκάλεσε οδήγησε σε πάρα πολλές ε, νέες ιδέες ε, για το πώς θα έπρεπε να αναδιαρθρωθεί και να αναδιαμορφωθεί ο χρηματοοικονομικός τομέας στην Ευρώπη ώστε να μην εξαρτάται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό τομέα. Όπως γνωρίζετε ε, ο τραπεζικός τομέας με 80-85% συμμετέχει οικονομικά στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ είναι 75-80% χρηματοδότησης από τις αγορές equity. Πρέπει πολύ περισσότερο από αυτές τις αγορές κεφαλαίων να δράσουμε στην Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Θα ήταν ίσως πολύ χρήσιμο αυτό για να μειωθεί ο κίνδυνος ο οποίος έγκυται και ε, επικεντρώνεται στον τραπεζικό τομέα μέσω αυτής της κατάστασης. Οι equity αγορές, equity, equity markets θα μπορούσαν να δώσουν μια τέτοια δυνατότητα για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, πράγμα που θα ήταν χρήσιμο. Στο άλλο άκρο της κλίμακας έχουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου έχουμε 27 εκατομμύρια ανέργους σε 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Αν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε όρους και προϋποθέσεις κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να απασχολήσει έναν άνεργο από το σύνολο των ανέργων, ε, τότε το πρόβλημα θα μπορούσε, να, ε, θα μπορούσε να επιληθεί. Αυτό είναι βέβαια η κασία. Όμως παρόλα αυτά χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κονδύλια υπό τη μορφή δανείων, πιστώσεων σίγουρα και με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αγορές ε, θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε τέτοια κονδύλια αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε όμως και νέα μέσα, νέα εργαλεία θα έλεγα αυτά είναι δύο από τα πιο σημαντικά στοιχεία ως ε, οδούς που θα μπορούσαμε να πορευτούμε, διάβλους που θα μπορούσαμε να διανύσουμε στην πορεία μας προς το μέλλον. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στο τραπέζι αλλά και πολλοί, πολλές σημαντικές ε, πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν και θα αναλυθούν. Προκλήσεις για την Ευρωζώνη τώρα που αναφέρατε. Φυσικά το κύριο κυριότερο πρόβλημα όχι μόνο για την Ευρωζώνη αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι η βάση ανάπτυξης, ε, ο ρυθμός ανάπτυξης ανάπτυξης που είναι μικρότερος από τον ρυθμό ανάπτυξης ε, στις οικονομίες των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των φθινοπορεινών συναντήσεων στην ε, Ουάσιγκτον <clears throat> δεν ασκήθηκαν επικρίσεις ε, και αυτό ήταν κάτι καινούριο στις συζητήσεις, στις διαβουλεύσεις. Όχι τόσο, δεν υπήρξαν επικρίσεις από το οικονομικό, θα έλεγα, στρατόπεδο, αλλά αυτό να το υπενθυμίσουμε, να το λάβουμε υπόψη σε σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν. Φαίνεται ότι αρχίζει η ανάπτυξη, η ανάκαμψη σε σχέση με εμά. και φαίνεται ότι υπάρχουν προοπτικές ε, να σταθεροποιηθεί με θετικό τρόπο. Πρέπει όμως να βελτιωθεί γενικά η χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Για μας η οικονομική ανάκαμψη είναι μία από τις προτεραιότητες ε, και πιστεύω ένα από τα κινήτρα για τα οποία προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενταχθούμε στην Ευρωζώνη είναι ότι πιστεύουμε πραγματικά στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Και ένα από τα επιχειρήματα υπέρ της Ευρωζώνης, ακριβώς για μένα όπως το βλέπω, είναι ότι η Ευρωζώνη καταφέρνει και κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα η ίδια αυτούσια αυτοτελώς έχει το δυναμικό και την ικανότητα να ξεπεράσει, να υπερβεί κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν πιστεύω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και για την Ευρωζώνη στο μέλλον. Εντάξει, αλλά η Ευρωζώνη είναι σε θέση να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις ε, δυσκολίες αυτοτελώς ε, η ίδια. Και όσον αφορά το FTT, το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, επετεύχθη κάποια σε τεχνικό επίπεδο πρόοδος, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, έχουμε διαδικασίες ε, διευρυμένης ε, ε, συνεργασίας, enhanced cooperation procedures, και σε σχέση με αυτές 11 χώρες για αυτή τη διαδικασία, για το μέλλον αυτού του τέλους χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τι θα γίνει τελικά, ποια έκβαση θα υπάρξει, νομίζω κατά την άνοιξη θα δούμε ποια θα είναι η πρόοδος. Κατά την άνοιξη 2014 οι συνάδελφοι της επόμενης προεδρίας, της ελληνικής προεδρίας θα μπορούν πολλά περισσότερα να σας αναφέρουν για αυτό το τέλος χρηματοοικονομικών συναντήσεων. Ευχαριστώ. Μια που ξεκινήσαμε στις 9.30 θα συνεχίσουμε με τον Υπουργό. Βάνα Μαλέτσι τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίζω και εγώ εδώ τον Υπουργό και τον συγχαίρω και εγώ για την επιτυχή Προεδρία που είχατε. Επιτυχή σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα επειδή ενισχύεται έτσι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, υπάρχουν νέες κατευθυντήριες γραμμές στη συνοχή, στη γεωργία, ε, θεματική συγκέντρωση, μακροπεριφερειακή στρατηγική κλπ. κλπ. Έχουμε συζητήσει εδώ επί μακρό την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κονδύλια, σε πιστώσεις. Το τονίσατε κι εσείς πόσο σημαντικό είναι. Βέβαια, η κατάσταση στις χώρες μέλη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ιδιαίτερα όταν Μιλάμε για τα επιτόκια, κάτι το οποίο οδηγεί σε ανισότητες μέσα στην ε, εσωτερική αγορά. Οι επιχειρήσεις δηλαδή δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όλες. Οπότε εσείς πώς σκέφτεστε ότι μπορεί να λυθεί αυτό και όχι μόνο μέσα στην Ευρωζώνη αλλά και εκτός Ευρωζώνης. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη. Κάτι σημαντικό που έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πώς θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι συστάσεις που έρχονται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή οι συστάσεις αυτές. Από την ανάλυση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, διαπιστώνουμε ότι μόνο δύο χώρες έχουν θέσει σε εφαρμογή τις συστάσεις και άλλες εν μέρη μόνο τις έχουν εφαρμόσει. Εσείς πώς βλέπετε το θέμα αυτό της εφαρμογής των συστάσεων. Γιατί δεν γίνεται, δεν είναι αρκετά σαφείς, συγκεκριμένες οι συστάσεις και τι θα έπρεπε να αλλάξει από αυτού. Τρίτη ερώτηση. Η εμπειρία που έχετε από τη δικιά σας χώρα στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Στις 21 Ιουνίου εσείς βγήκατε από τη διαδικασία αυτή υπερβολικού ελλείμματος. Ε, προχωρήσατε σε μέτρα όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες. Σχετικά με τις δαπάνες, ένα μέτρο ήταν η μείωση των μεταφορών στον πυλώνα για τις συντάξεις. Εσείς στη Λιθωνία έχετε σκεφτεί το θέμα της κατάργησης του δεύτερου πυλώνα και πώς αξιολογείτε την μείωση των μεταφορών αυτών στο έλλειμμα. Πώς βοήθησε αυτό για την μείωση του γενικού ελλείμματος. Πρόεδρος. Προεδρεύων. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Κοιτάξτε, έχω μπερδευτεί λίγο, γιατί εδώ βρίσκομαι ως ε, πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ. Οπότε ίσως δεν θα ήταν σωστό να συζητήσω εδώ μαζί σας θέματα εσωτερικά της Λιθουανίας. Ζητώ συγγνώμη, αν θέλετε, μπορούμε σε προσωπικό επίπεδο διμερός να το συζητήσουμε, αλλά δεν θα ήθελα να το συζητήσω αυτό εδώ δημοσίως. Τώρα για την πρώτη σας ερώτηση, πολύ σημαντική η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Τα επιτόκια φυσικά και αποτελούν σημαντικό παράγοντα και μερικές φορές εμποδίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν χρηματοδότηση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας, ακόμα πιο σημαντικός. Και αυτό είναι η δυνατότητα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από τι τράπεζε οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλέ φορέ οι τράπεζε δεν θέλουν να αναλάβουν κίνδυνο. Οπότε με κανένα επιτόκιο δεν δανείζουν χρήματα αν δεν είναι σίγουρες ότι η επιχείρησή σας θα τα πάει καλά. Εδώ όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τόσο σημαντικό στοιχείο της οικονομίας μας που πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν ε, τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην ε, νιώθουν οι τράπεζες αυτό το κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζουν να συμπεριλάβουν μέτρα τα οποία θα μειώσουν τον κίνδυνο αυτό. Αυτά τα μέτρα συνδυάζονται με διαρθρωτική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό Οπότε, εφόσον υπάρχουν εγγύησει ή εν πάση περιπτώσει μειωθεί ο κίνδυνος, τουλάχιστον έτσι τον βλέπει ιδιωτικό τομέα, τότε θα διευκολυνθεί η χρηματοδότηση αυτή. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε είναι να φροντίσουμε για τις νομικές διατάξεις τους κανονισμούς για τη συνοχή, ώστε οι χώρες μέλη να μπορούν από μόνες τους να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά. Στη Λιθουανία τα χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά. Ένα από τα σλόγγαν που ήταν ιδιαίτερα επιτυχές αλλά και σημαντικό στη συνάντηση στο Βίλνιους με τους Υπουργούς Συνοχής ήταν για τα ευρωπαϊκά χρήματα. Το εξή. Καλύτερα επενδύσεις παρά καλές δαπάνες. Οποιαδήποτε επένδυση είναι καλύτερη από την οποιαδήποτε καλή δαπάνη. Πολύ σημαντικό αυτό. Στις συζητήσεις που θα έχουν οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων σε λίγες μέρες, εκεί θα γίνει αξιολόγηση του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Φυσικά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στις συστάσεις. Υπάρχουν γενικές συστάσεις που αφορούν όλες τις χώρες. Άλλες είναι πολύ συγκεκριμένες για επιμέρους χώρες. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται και τα δύο. Και οι γενικές συστάσεις και οι ειδικέ συστάσεις ανά χώρα. Αλλά πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική ανάλυση για το πώς οι συστάσεις αυτές εφαρμόζονται στην κάθε χώρα. αν έχετε μία σύσταση, την επόμενη χρονιά αυτή τίθεται σε εφαρμογή. Αλλά στην πράξη δύσκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν συστάσεις που επαναλαμβάνονται για χρόνια για μία χώρα. Ξανά και ξανά. Και υπάρχουν θέματα για τα οποία έτσι αλλιώς και η πρόοδο είναι κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αν υπάρχει κάποια πρόοδο στην απασχόληση, για παράδειγμα στην αντιμετώπιση του ελλείμματος. Αυτό είναι ήδη θετικό. Νομίζω πάντως ότι μετά το Εαρινό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Πρόεδρος, εγώ θέλω όταν είπα ότι έχουμε ακόμα χρόνο να ολοκληρώσω τον κατάλογο ομιλητών για ερωτήσεις, όχι για να προσθέσω κι άλλους. Ε, Σίμωνα, τους σοσιαλιστές. Μάλιστα, Πρόεδρε, και εγώ θυμάμαι τις πρώτες μας συζητήσεις ακριβώς εδώ, ακριβώς εκεί που κάθεστε, μετά από την πρώτη συζήτηση στο, στην ΕΚΟΝ συζητήσαμε αν υπάρχει καν κάποια ευκαιρία το τρίτο τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία να την ολοκληρώσουμε, την ασφάλεια καταθέσεων. Και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ θερμά για την απίστευτη αφοσίωση, προσπάθειες εξαιρετικές και την τόσο επικοδομητική συνεργασία που είχαμε και με τους συνεργάτες σας με το Ευρωκοινοβούλιο συνολικά. Εγώ ευελπιστώ απόλυτα, είμαι αισιόδοξο ότι έχουμε ευκαιρίες αυτή την ε, αυτό το θέμα ε, παρότι έχουμε διαφορές απόψεων απόψε στον τριμερή διάλογο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Άξιζε σίγουρα η πορεία που διανύσαμε. Πολλά προβλήματα τα αντιμετωπίσαμε και τα επιλύσαμε που κανείς δεν θα το πίστευε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα διανύαμε τόσο μεγάλη πορεία. Χαίρομαι και εγώ και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε απόψε το τελευταίο μέρος της πορείας να το καλύψουμε απόψε. Ευχαριστώ για αυτόν τον τρόπο συνεργασίας που μέχρι σήμερα στη θητεία μου ποτέ δεν το έζησα αυτό, δεν το βίωσα Έχω μία ερώτηση που με προβληματίζει κάπω, ε, βλέποντας όχι μόνο τις καθημερινές, ε, τα όσα τεκταίνονται καθημερινά, αλλά και την προοπτική στο μέλλον. Και για αυτό το χαρτοφυλάκιο, όλο και για άλλα θέματα. Βλέπω ότι ο ρόλος που εμείς στην ΕΠΑ θέλαμε να δώσουμε ως ε, αρμοδιότητες όταν δημιουργήθηκε αυτό και πώς εξελίχθηκε επ' αυτού ότι έχουμε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας σήμερα. Αν σκεφτώ και θυμηθώ για την ε, δημιουργία της ε, εποπτικής αρχής, ε, τι, ποιες ελπίδες και προσδοκίες είχαμε αρχικά και βλέποντας τώρα ότι με κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται στο Συμβούλιο κάθε κείμενο, κάθε πρόταση εγώ τουλάχιστον για το κείμενο επί του οποίου εργάζομαι εγώ μπορώ να το διαπιστώσω αυτό και να το δω για την ασφάλεια καταθέσεων. Αποδυναμώνονται οι προτάσεις οι αρμοδιότητες. Έχουμε ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που σε σχέση με τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου μειώνονται ή ας το πω έτσι αποδυναμώνονται. Εδώ έχουμε και την παρέμβαση και των κρατών μελών. Όλα αυτά με ανησυχούν. Ποτέ δεν φανταζόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Εποπτείας ε, θα ήταν ένα ενδιαφέρον σώμα διαβούλευσης. Εμείς πιστεύουμε θα έπρεπε να είναι μια αρχή με κύρος και αρμοδιότητες. Πώς βλέπετε εσείς ε, την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ε, ε, Εποπτικής Αρχής Τραπεζών. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα Πρέπει επίσης και εγώ να σας ευχαριστήσω εσάς και πάλι για αυτή την πάρα πολύ παραγωγική συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου της Προεδρίας μας. Υπό το δικό μου πρίσμα ήταν μια εξαιρετική συνεργασία, ιδιαίτερα με την Οικονομική Νομισματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα, αφορώντας το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, είναι μια πολύ σημαντική αρχή αυτός ο θεσμός. Είναι, δεν είναι όμως ε, ασυνήθιστο να μεταθέτονται αρμοδιότητες και εξουσίες ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων μετά την συγκρότηση και ίδρυσή τους ε, όταν έχει επιτευχθεί κάποια πρώτη φάση και προχωρούμε στον τραπεζικό τομέα και για την ρύθμιση του τραπεζικού τομέα ιδιαίτερα όχι μόνο για τις χρηματοοικονομικές αγορές σφαιρικά αλλά και για τον τραπεζικό τομέα <clears throat> δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε ένα συγκεκριμένο τελεσίδικο αποτέλεσμα. Μετά τη δημιουργία και έναρξη σε λειτουργία και ισχύ του ενιαίου τραπεζικού εποπτικού μηχανισμού, τώρα από σε, σχέση με τα ε, stress tests, τις δοκιμές, ε, δοκιμασίες ε, φέτος και στη συνέχεια όταν θα αρχίσει να ισχύει ο ενιαίος εποπτικός τραπεζικός μηχανισμός, έχοντας ήδη καθορίσει το θέμα του, της Προεδρίας και της Αρμοδιότητας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προγραμματίζεται και σχεδιάζεται το έργο αυτό. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει κατά το επόμενο έτος. Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους, κατά το Δεκέμβριο 2014, μετά από ένα έτος, θα είναι πολύ σαφέστερο ποιος θα βρίσκεται πού, ποιες αρμοδιότητες θα έχει, ποιο θα είναι το καθήκον του και το έργο του και οι αρμοδιότητες του. Είναι θα έλεγα ομαλό και κανονικό ότι είναι κάπως μετέωρα τα πράγματα και ρευστά αυτή τη στιγμή. Θα καθοριστούν όμως ε, με την πάροδο του χρόνου. Τελική ερώτηση. Ο κύριος Μπαντίνη παρακαλώ. Ε, ναι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Υπουργέ για την εξαιρετική εργασία που έχετε κάνει, για τις πολύ σημαντικές επιτυχίες της Προεδρίας σας. Συγχαρητήρια λοιπόν προς τον Υπουργό τον κύριο Σάτζιους για τις σημαντικές αυτές επιτυχίες της Λιθουανικής Προεδρίας. Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των επιτυχιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, θα ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας όσον αφορά τα αποτελέσματα που, έχουμε, που έχει πετύχει η ίδια η Λιθουανία κατά τη διάρκεια της προεδρίας αυτής. θεωρείται γενικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υποφεληθεί από την δική σας την συμμετοχή. Ενδεχομένως από συμβολικής πλευράς η Λιθουανία έδωσε πολύ περισσότερα από όσα τελικά πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας συγχαρώ επίσης και για τα μέτρα τα οποία λάβατε στον τομέα της αγοράς, στον τομέα των αγορών Σας ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ για τα πολύ ωραία δώρα τα οποία μας δώσατε, αυτές οι καταπληκτικές ε, γραβάτες. Εγώ τη δική μου την άφησα στο σπίτι μου, στην Κροατία. Νομίζω πάντως ότι θα μου πήγαινε πάρα πολύ αν τη φορούσα τη γραβάτα αυτή σήμερα. Σάρα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ακούσω καλύτερη ερώτηση για το τέλος. Πραγματικά θα μπορούσα να ονειρευτεί καλύτερη ερώτηση και καλύτερα σχόλιο. Ναι, αλλά λυπάμαι ο κύριος Λάγκε πρέπει να κάνει τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι χαίρομαι πάρα πολύ που την 1η Ιουλίου η Λιθουανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά και η Κροατία προσχώρησε εκείνη την ημερομηνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγινε το 28ο μέρος της Ένωσης. Απαντώντας λοιπόν στη δική σας την ερώτηση θα έλεγα το εξής. Όπως και σε μια οικογένεια Ποτέ δεν θα ρωτούσε κανείς κάποιον μια ερώτηση, ένα μέλος οικογένειας, αν έχει αποφεληθεί ή όχι από το άλλο μέλος. Λειτουργούμε σαν οικογένεια και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η εμπειρία η οποία είχα εγώ στην πολιτική μου ζωή ήταν η καλύτερη δυνατή, η εργασία μου αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι κατάφερα πραγματικά να βιώσω αυτή την πραγματική ζωντανή οικογένεια που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πρόκειτο για μια στήρα τυπική συνεργασία μεταξύ κυρίαρχων απομονωμένων κρατών μελών όπως πολλές φορές βλέπουμε σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μια πραγματική οικογένεια και το οικογενειακό αυτό συνέστημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά και γενικότερα για τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ερώτησή σας και συμφωνώ μαζί σας ότι η γραβάτα είναι καταπληκτική. Η τελευταία όμως τώρα ερώτηση πραγματικά από τον κύριο Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου την εντύπωση που ανέφεραν οι συνάδελφοι να την επιβεβαιώσω. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας αυτό το εξάμεινο πετύχατε εξαιρετικά ειρηνική σύναψη συμφωνιών και ολοκλήρωση χαρτοφυλακίων. Είναι μια από τι σπάνιε στιγμέ που στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί κανεί ε, ειλικρινά να εκφράσει τέτοιου επένου. Μια άλλη ερώτηση. Είπατε ότι ω Προεδρεύον του ΕΚΟΦΗΝ είσαστε παρόν. Σήμερα το απόγευμα, γύρω στι 3 το απόγευμα, το μέλο ε, ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κύριο Άσμουσεν, θα διοριστεί υφυπουργό στη νέα Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τη Γερμανία. Στη συνέχεια, ο κύριο Ντράγκη, ο οποίο ήταν εδώ εχθέ Δευτέρα, θα αποστείλει μια επιστολή στην, ε, ε, για την αναπλήρωση του κυρίου Άσμουσεν στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση που θα χειρεύσει δηλαδή μετά την αποχώρηση του Άσμουσεν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα παρουσιαστεί ίσω κατά τη διάρκεια αυτού του ΕΚΟΦΗΝ αυτή η επιστολή και έτσι θα ξεκινήσει μια διαδικασία για την πλήρωση τη ε, θέση του μέλου του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που η θέση του χειρεύει τώρα. Τώρα, Πάντα επανειλημμένα είχαμε συζητήσει ότι ο αριθμός των γυναικών στο Διοικητικό Συμβουλίο είναι υπερβολικά μικρός. Αυτό οδήγησε στο ότι έπρεπε να υπάρξει αναμονή ενός ε, εξαμήνου για να μπορέσει το πράγμα να αλλάξει. Τώρα ε, διορίστηκε ο κύριος Άσμουσεν μετά από συμφωνία, μετά από γερμανική πρόταση στη θέση αυτή. Δεν πέρασαν ούτε δύο χρόνια. Το θεωρείται σωστό να γίνει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντράγκη. Και δεύτερον, να έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης για αυτή τη θέση η Γερμανία, μια ε, είχε ε, υποβληθεί αυτή η πρόταση αρχικά είναι μια επίκαιρη ερώτηση Υπουργέ. Ίσως δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να απαντήσετε. Αλλά θα βρεθεί μπροστά σας το ερώτημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Uh, uh, Ο Υπουργό. Φυσικά σε ευχαριστώ για την ερώτηση που διατυπώσατε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Γιώργο Γκάσμουσεν με τον οποίο συνεργαστήκαμε έντονα κατά τη διάρκεια των ΕΚΟΦΗΝ των Συμβουλίων. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στην επόμενη πολιτική του σταδιοδρομία, διότι δεν ήταν πολιτικό διορισμό στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εν παρόδο είναι σοσιαλδημοκράτη όπω και εγώ. Τώρα, όσον αφορά τι διαδικασίε αυτέ τι οποίε αναφερθήκατε, φοβούμαι ότι δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τη συγκεκριμένη σα ερώτηση αυτή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της εντολής ε, θέσαμε έγιναν πολλά ρεκόρ ως επιδόσεις ε, σε σχέση με τους τριμερείς ε, διαλόγους, νομοθετικό έργο το οποίο επετεύθη τώρα και σε σχέση και με τον αριθμό ατόμων και τον διορισμό τους ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ας ελπίσουμε ότι ο, δεν θα συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η ανακύκλωση. Τώρα, ελπίζουμε ότι αυτό σίγουρα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα υπάρξουν αυτές οι επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε για τις διεξοδικές σας απαντήσεις και φυσικά και όλους τους συνεργάτες σας για αυτή τη συνεργασία. Συμμετέχω σε όλους τους τριμερείς διαλόγους και γνωρίζω ότι έχουν πραγματικά ότι έγινε μια εξαιρετική δουλειά και από πλευράς της χώρας και της Προεδρίας σας αυτό μπορεί να σας κάνει υπερήφανος. Σάρον ε, παρεμβαίνει ο Πρόεδρος. Απλά δύο τελευταία λόγια να πω. Θα ήθελα επίσης να μου επιτρέψετε παρισφρέοντας τη διαδικασία αυτή όχι απλά και μόνο παραδοσιακά να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες προς την Σάρων ατομικά για αυτόν τον πολύ γόνιμο, πολύ ενδιαφέρουσα και ενθαρρυντική συνεργασία. Θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω Σάρων Μπόλς. Θα σε ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Μπόλς. Τώρα θα δώσω την προεδρία. έχω και δωράκι. Μάλιστα. Για σας που δεν το γνωρίζετε συμμεριζόμαστε ένα παρόμοιο προηγούμενο ε, θα έλεγα ε, χαρακτηριστικό και γι' αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή προεδρία ιδιαίτερα αυτή. Τώρα θα δώσω τον, την προεδρία στον Παύλο. Ναι, έχεις τώρα μπορείς να προεδρεύσεις Παύλο. Eh, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες. Για το θέμα αυτό είμαι εγώ εισηγητής. Πρόκειται για κοινή συζήτηση που συμπεριλαμβάνει και τις υπηρεσίες πληρωμών. Για το θέμα αυτό είναι εισηγητής ο κύριος Φέιο. Λοιπόν, θα παρουσιάσω την έκθεσή μου, μετά ο κύριος Φέιο θα παρουσιάσει τη δικιά του έκθεση και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους κοιόδες εισηγητές και για τις δύο αυτές εκθέσεις. Οπότε, σας παρουσιάζω τη δικιά μου έκθεση. Πρώτα απ' όλα. Εντάξει, είναι περίεργο να προεδρεύει κανεί τη συνεδρίαση όπου παρουσιάζει την έκθεσή του, αλλά τι Λοιπόν, κύριο στόχο τη έκθεση αυτή είναι να πετύχουμε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, τη διαφάνεια. Να πετύχουμε δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα πληρωμών που να διέπεται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αν το πετύχουμε αυτό θα είναι ήδη κάτι πολύ καλό. Πολλοί επικρίνουν το θέμα των διατραπεζικών ε, προμηθειών που δεν είναι ίδιες και που έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τελικά το κόστος της κάρτας πληρωμής. Οπότε, αν το πετύχουμε, βέβαια έχω τις αμφιβολίες μου, δεν θα έπρεπε. Αλλά αν μη τι άλλο, ο στόχος της ε, διαφάνειας είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε. Τότε οι καταναλωτές θα ξέρουν τι ακριβώς πληρώνουν κάθε φορά που χρησιμοποιούν την τραπεζική τους κάρτα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Και αυτό είναι κεφαλαιόδου σημασία, όχι μόνο για την έκθεση αυτή, αλλά για οποιαδήποτε νομοθετική έκθεση που παρουσιάζουμε. Κατά τη γνώμη μου πάντα πρέπει να έχουμε σαν στόχο την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Τρίτος στόχος είναι άπαξ και αρχίσει να ισχύει η έκθεση αυτή και η έκθεση του κ. Φέιο, οι διάφορες επιχειρήσεις να έχουν κίνητρα προκειμένου να προχωρούν στην καινοτομία. Και αυτό είναι κεφαλαιόδου σημασία πρέπει να προχωράμε με καινοτομία μέσα στα συστήματα πληρωμών. Και ο τελευταίος μας στόχος, εξίσου σημαντικός, είναι να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών. Οπότε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει βασίσει τις προτάσεις της σε μια στέρεα, γερή μελέτη ώστε να αποδεικνύονται τα ωφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση πιο προσεκτική και με περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε χώρα μέλος. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, το επίπεδο που χρησιμοποιείται η πληρωμή με κάρτα στις χώρες μέλη διαφέρει. στόχος της μελέτης αυτής θα ήταν να μην έχουμε αντίθετε επιπτώσεις από αυτές που επιθυμούμε να έχουμε από την χρήση των ε, καρτών αυτών πλήρωμή. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η νέα νομοθεσία σε όλες τις χώρε μέλη θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Θα επιτευχθεί δηλαδή η αύξηση της χρήσης των πληρωμών με πιστοτικές κάρτες. Τα πιο επίμαχα θέματα τώρα θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί σας, να ακούσω και τους κοιόδης εισηγητές και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Εγώ στην έκθεσή μου αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι να υπογραμμίσω τα θέματα αυτά που πιστεύω ότι είναι πιο επίμαχα, να εντοπίσω τα ζητήματα για τα οποία πιστεύω πρέπει να βρούμε μια καλύτερη λύση. Γι' αυτό και προτείνω στην έκθεσή μου μια λύση όμως χρόνος είμαι ανοιχτή απέναντι στους ε, άλλους σκιώδες ηγητές και την Κομισιόν για να προσπαθήσω να βρω εναλλακτικέ λύσεις. Σε σχέση με το άρθρο 1, πεδίο εφαρμογή. η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκλεί από τα, τριμερή συστήματα από την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με τα όρια των διατραπεζικών προμηθειών και από τις διατάξεις του άρθρου 7 σχετικά με τον διαχωρισμό των καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση αυτή πρέπει να προσφέρει ίσους όρους στον ανταγωνισμό για όλα τα συστήματα και των τριμερών και των τετραμερών αλλά και των διαφόρων φορέων επεξεργασίας. Όσον αφορά τώρα τα άρθρα 3 και 4 διατραπεζικές προμήθειες που αποτελούν και την καρδιά της έκθεσης αυτής. Εγώ κρατώ την πρόταση της Επιτροπής, αλλά θεωρώ συγχρόνως ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των ορίων που προβλέπονται. Να γίνει δηλαδή μια περισσότερο σε βάθος αξιολόγηση προηγουμένως, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στα κράτη-μέλη όπου οι αγορές των, ε, με τα μέσα αυτά πληρωμής είναι πιο αναπτυγμένες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διατραπεζικές προμήθειες δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε μικρότερη χρήση των καρτών αυτών. Οι διατραπεζικές προμήθειες δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδι σε επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων πληρωμών και στις χώρες εκείνες όπου οι κάρτες αυτές δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ όπως άλλες. Και δεν θα πρέπει να σημαίνει λιγότερες επενδύσεις για την καινοτομία. Προς το παρόν αποφάσισα την εισαγωγή κάποιες ελαστικότητας στις διατραπεζικές προμήθειες, ώστε να γίνεται στάθμιση ανάλογα με τα απόλυτα όρια τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι ίσως αυτό να μην είναι η τέλεια λύση. Είναι όμως η λύση που προτείνω, αλλά όπως σας είπα είμαι διατεθειμένος να ακούσω και εναλλακτικέ λύσεις για να πετύχουμε τον επιθυμητό στόχο. Η πρότασή μου θα επιτρέψει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τομείς που έχουν διαφορετικά, ε, διαφορετικές τραπεζικές προμήθειες ή διαφορετικούς ε, κινδύνους που λοχεύουν, ώστε οι πληρωμές να είναι πιο ασφαλείς. Συνεχίζουμε να συζητάμε και να προβληματιζόμαστε απέναντι σε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Εγώ αυτά είχα να πω και θέλω να ακούσω τους συναδέρφους τώρα για τα σημεία που θεωρούν πιο σημαντικά. Αλλά έρχομαι και στο άρθρο 2 που αναφέρεται στις διασυνοριακές συναλλαγές, τον ορισμό δηλαδή. Ο ορισμός αυτός με κάνει να έχω κάποιες αμφιβολίες για το τι επιπτώσεις θα έχει αυτός ο νέος ορισμός και μήπως δημιουργηθούν ανισορροπίες ανάμεσα στις εσωτερικές αγορές και τις άλλες. Στις εσωτερικές συναλλαγές ακολουθούμε τον παλιό ορισμό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν επηρεάζονται στην μεταβατική περίοδο των 22 μηνών οι εσωτερικές αυτές αγορές. Πάντως το άρθρο 2 που αναφέρεται στην πληρωμή με χρεωστικές και πιστοτικές κάρτες. Οι ορισμοί που εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πληρωμές με χρεωστικές και πιστοτικές κάρτες επιδέχονται βελτίωση. Και εδώ θέλω και την άποψη των υπολείπων για να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε ορισμούς που να είναι σαφείς και εφαρμόσιμοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα τη διάκριση ανάμεσα στα συστήματα και τους φορείς επεξεργασίας. Στο άρθρο 7 Ίσως είναι υπερβολικό να πετούμε την διάκριση, το διαχωρισμό των καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας ανάλογα με την ε, ε, φυσική τους, την νομική τους, ε, το νομικό πρόσωπο. Έχω κάποιες αμφιβολίες εδώ. Θα πρέπει να είναι λειτουργική η διάκριση και να διασφαλίζουμε ότι η παρουσίαση των υπηρεσιών δεν θα επηρεάζει την αποδοχή όχι άλλων υπηρεσιών. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση γεωγραφικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούν τα συστήματα πληρωμής. Οι φορείς επεξεργασίας της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι το σύστημά τους τεχνολογικά είναι λειτουργικό και συνδυάζεται και είναι συμβατό με τα άλλα συστήματα που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος που επιτρέπει στους διάφορους φορείς να προσαρμοστούν. Όσον αφορά το άρθρο 8, όσον αφορά την επιλογή δηλαδή των λειτουργιών. Εδώ μπορεί να υπάρξουν διαφορετικά αποτελέσματα από τα επιθυμητά, δηλαδή να είναι τελικά πιο δύσκολο να υπάρχουν λιγότερα κίνητρα προκειμένου να θέλει κανείς να πληρώσει με ε, κάρτα πληρωμής. Είτε όταν πρόκειται για προεπιλογή και είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να επιλέξει τα διάφορα σήματα, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και επιπλοκές για τους χρήστες. Μπορεί να κάνω λάθος και να μπερδευτούν τη στιγμή της πληρωμής. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για τις κάρτες, έτσι. Αν πρόκειται για τα κινητά ή άλλο τρόπο πληρωμής, τότε είναι διαφορετικό. Αλλιώ είναι αυτό που ονομάζουμε το πλαστικό χρήμα και αλλιώ είναι οι πληρωμέ που γίνονται με άλλου είδου μέσα, όπω είναι η επαφή ή το κινητό. Ο στόχος τελικά πρέπει να είναι να διευκολύνουμε το, τη ζωή στους καταναλωτές και γι' αυτό αυτό είναι ο στόχος που πρέπει να καθοριστεί ή και να αξιολογηθούν οι διαφορετικές δυνατότητες που αναφέρονται στο θέμα αυτό σε σχέση με το άρθρο 10 δηλαδή που θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη ε, όλες οι κάρτες ε, δηλαδή υποχρέωση αποδοχής όλων των καρτών θεωρώ ότι ίσως αυτός ήταν ο πιο σημαντικός μηχανισμός για την χρήση των καρτών ως μέσο πληρωμής. Αυτή η πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει σαν συνέπεια οι κατανάλωτες να δουν ότι οι κάρτες τους δεν γίνονται δεκτές κατά τη στιγμή που επιθυμούν να πληρώσουν με αυτές διότι όταν υπάρχει σε κάποιο μαγαζί μια μάρκα και μετά μια ε, κάρτα πιστοτική και δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί με αυτή την πιστοτική κάρτα ο λογαριασμός δημιουργείται απουσία εμπιστοσύνης τουλάχιστον για τους καταναλωτές και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και να είναι πιο δυσχερή η πληρωμή με τραπεζικέ κάρτε και να μην επιτυγχάνεται η επίτευξη μέσω αυτή τη νομοθεσία τη ευρύτερη χρήση των τραπεζικών καρτών. Γι' αυτό αν αληθεύει λοιπόν ότι αυτό είναι ο στόχο αυτής της πρόταση. είμαι ανοιχτό να αναζητήσουμε ενδιάμεσε προτάσει και λύσει. με έναν ενιαίο μοναδικό στόχο. Ο όταν θα μπαίνει σε ένα μαγαζί να έχει την δυνατότητα και τη βεβαιότητα, να έχει την βεβαιότητα σε σχέση με τον λογότυπο της ε, κάρτας του για να μην υπάρχει ε, το ε, πρόβλημα, να μην δημιουργείται πρόβλημα στην πληρωμή με κάρτα. Αυτά είναι τα προβλήματα που είδα και εντόπισα και αναφέρω στην έκθεση που έχω την τιμή να είμαι εισηγητής για αυτήν. Αυτές οι λύσεις, αυτές οι λύσεις δεν είναι αμετακίνητες και ε, δεδομένες ως θέσφατα. Είμαι ε, πρόθυμος να αναζητήσω λύσεις με τους γιώδεις εισηγητές και με όλους όσους εμπλακούν σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική θητεία στη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για την υπομονή για τις επεξηγήσεις που σας έδωσα. Δίνω τον λόγο στον συνάδελφο Διego Φεγιό και πρέπει να πω ότι ήταν τιμή να ε, μπορώ να συνεργαστώ μαζί του και θα ανοίξει η συζήτηση μετά με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Διόγκο, στον τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ από πλευράς μου με το τελευταίο λέγοντας ότι οι αρχικές εργασίες σε σχέση με αυτά τα δύο, με αυτά τα θέματα των δύο εκθέσεων καταδεικνύει ότι ήταν δυνατόν οι δύο εισηγητές και οι βοηθοί τους να συνεργαστούν σε μια ομάδα συνολικά και αυτό ήταν πολύ θετικό. Παρόλη τη διαφορά μεταξύ κανονισμού και οδηγίας υπάρχει λόγος ύπαρξης για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων σε μια δέσμη μέτρων, σε ένα ενιαίο πεδίο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας αυτή την πτυχή. Οι σχεδόν 20 τόσες τροπολογίες που είχα την ευκαιρία ήδη να παρουσιάσω για αυτή την έκθεση ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα πρώτο βήμα που θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με ε, την εργασία μας. Δεν είναι σίγουρα μια τελική διατύπωση, καθοριστική τελεσίδικη ε, διατύπωση. Ανταποκρίνονται στις ιδέες και απόψεις που έχω για τη διαμόρφωση αυτού του συνόλου θεμάτων σύμφωνα <clears throat> με εκείνα τα οποία θεωρήθηκαν από μένα τα κυριότερα θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν και να ρυθμιστούν από αυτή την οδηγία. Η ασφάλεια, η δημιουργία εμπιστοσύνη, η απλούστευση, ο απλό χαρακτήρα, ο ανταγωνισμό επίση, η ενημέρωση και πληροφόρηση και η ικανότητα προσαρμογών προσαρμογών σε σχέση με αυτές τις νομοθεσίες, με αυτά τα νομοθετικά ε, πλαίσια για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Και το έργο πέρασε μέσα από δεκάδες συνεδριάσεις και με διάφορους εμπλεκόμενους στην αγορά. Ευχαριστούμε επίσης όχι μόνο για αυτές τις συνεδριάσεις και επαφές αλλά και για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν και που ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις προτάσεις που ε, υποβάλλω με πρόθεση να είναι ισορροπημένες οι προτάσεις αυτές και για να δοθούν αποτελεσματικές απαντήσεις στις ανάγκες των αγορών. Πρέπει επίσης να προσθέσω σαν ένα άλλο στοιχείο ότι με ικανοποίηση, γενικότερη ικανοποίηση αποκόμισα ε, θετικές εντυπώσεις σε σχέση με το ε, κείμενο, σε σχέση με την υφιστάμενη νομική ρύθμιση και τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει. Σε σχέση με τις τροπολογίες, τροποποιήσεις που υποβάλλονται σε σχέση με την αρχική πρόταση, για να μην μακρηγορήσω και σας επιβαρύνω και να μην είμαι εξαντλητικός θα επικεντρωθώ σε τέσσερα κυριότερα θέματα. Το πρώτο από αυτά ε, αφορά τα τέλη, charges. Υιοθέτησα μία θέση στην οποία θεωρούσα ότι οι ιδιομορφίες πρέπει να καλυφθούν και οι διαφορές ε, σε σχέση με τις εθνικές αγορές και πραγματικά υπάρχουν διαφορές και υπάρχει κατακαιρματισμός σε σχέση με τις απόψεις για αυτό το θέμα. Αφήνω στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την ελευθερία, διακριτική ελευθερία, να επιλέξουν την ίσπραξη τελών, surcharges, ή να την επιτρέψουν. Πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο που το κόστος που εδώ σε σχέση με την τιμή θα πρέπει να αναφέρεται το τέλος αυτό θα πρέπει να είναι η τιμή την οποία θα επομίζεται ο εμπορευόμενος, ο έμπορος σε σχέση με τη χρήση του μέσου πληρωμής ε, της κάρτας. Το δεύτερο σημείο αφορά τα TPPs σε σχέση με την συνοδεία, συνόδευση που πρέπει να υπάρξει, παρακολούθηση σε σχέση με τις ανάγκες των αγορών. Αυτά ήδη λειτουργούν και βρίσκονται σε μια αγορά που βρίσκονται, βρίσκεται εκτός ρυθμιστικού πλαισίου και γι' αυτό είναι σημαντικό να ενταχθεί, να εμπλαισιωθεί μέσα στο πλαίσιο των πληρωμών αυτών και μέσα σε αυτή την εμπλαισίωση, την ένταξη να θεσπιστούν κανόνες και διατάξεις διατάξεις και κανονισμοί για την λειτουργία τους και για τις ε, ε, συναλλαγές αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτή τη λογική, δηλαδή να υπάρχει ένα ενιαίο λειτουργικό πλαίσιο για αυτές τις λειτουργίες και να υπάρχει μια κανονική λειτουργία της αγοράς, καταλήγουμε στα εξής μέτρα. Υποχρεωτική καταχώρηση αυτών των ε, εμπλεκόμενων από πλευρά των αρμόδιων αρχών και ε, πλήρης ένταξη σε σχέση με τους, τον αγοραστή και την τράπεζα του αγοραστή μέσω της σωστής ετικετοποίησης ώστε να υπάρχει η έγκριση για την πρόσβαση, έγκαιρη πρόσβαση στον λογαριασμό, τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή και περιορισμός της ε, ε, διαθέσιμης πληροφόρησης ε, όσον αφορά αυτή την προσπελασιμότητα. Θα πρέπει απλά και μόνο να διατίθεται πληροφόρηση σε σχέση με την ύπαρξη κεφαλαίων που θα υπαρκούν, δηλαδή ρευστών, στο λογαριασμό που θα υπαρκούν για την αγορά αυτή. Η επόμενη πτυχή αφορά την ευθύνη, την υπευθυνότητα. Και για τις περιπτώσεις λοιπόν εκείνες στις οποίες υπάρχει μια χρέωστη πληρωμή που γίνεται σε σχέση με μια συναλλαγή όπου εμπλέκεται μια τέτοια λειτουργία με χρήση κάρτας είναι υποχρεωτική η επιστροφή, η ανάκτηση αυτών των χρημάτων. Και είναι θέμα του ΤΠΠ να μπορέσει να εφαρμόσει την πρόταση αυτή. Το τρίτο μεγάλο, ε, η κατηγορία τροποποιήσεων αφορά τα θέματα ασφάλειας. Όπως είναι προφανές, αυτά τα συστήματα πληρωμών πρέπει να έχουν μια ασφάλεια που θα τα καλύπτει, διότι η ασφάλεια εκείνη είναι που θα δημιουργήσει το κλίμα εμπιστοσύνης για τις πληρωμές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν έχουμε εδώ συναλλαγές που είναι διασυνοριακές και συναλλαγές που εμπλέκουν για παράδειγμα ηλεκτρονικά μέσα και όπου δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζει ο αγοραστής άμεσα τον πολιτή. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει η ασφάλεια, η διασφάλιση του πλαισίου ασφάλειας όλα τα συστήματα και διατάξεις να προβλέπονται και να μπορούν να λειτουργήσουν ώστε εκείνος που αγοράζει να πληρώνει μόνο για το αντίτιμο της συναλλαγής της αγοράς χωρίς να υπάρχουν ε, ε περιτές επιβαρύνσεις για πληρωμή ή αχρέωστες ε, ε, μη δικαιολογημένες πληρωμές εδώ σε σχέση με μη δικαιολογημένε πληρωμέ και στο πλαίσιο των απατών που μπορεί να συμβαίνουν, υπάρχει μεγάλο περιθώριο πιστοδρόμηση αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα λοιπόν ώστε η περίπτωση απάτης να αποκλείεται και να, να μην ε, μπορεί να υπάρξει. Έτσι ήμουνα υπέρ του εξή ύπαρξη δημόσιων μητρώων και καταλόγων που θα είναι καθολικά προσπελάσιμα αυτά τα μητρώα σε σχέση με τις ε, ε, εταιρείες που θα είναι ε, διαπιστευμένες. Και σε σχέση με τράπεζες, όταν θα υπάρχει μια αδικαιολόγητη παρέμβαση σε σχέση με τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορεί να παγώσει τις, ε, τις συναλλαγές με, ένα τέτοιο ε, πάροχο υπηρεσίας η τράπεζα. Εδώ η δυνατότητα λοιπόν μπορεί να οδηγήσει στο να αποσυρθεί η έγκριση λειτουργίας σε κάποιες εταιρείες στην, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν σημειωθούν τέτοια ε, συμβάντα. Αυτές οι προτάσεις που υποβάλλω είναι προφανώς προτάσεις οι οποίες είναι ανοιχτές στη διαπραγμάτευση και τροποποίηση. Πέρα όμως από τις τροπολογίες που κατέθεσα στο ΠΣΤ1 έχω και κάποια καινοτόμα στοιχεία τα οποία έχουμε μπροστά μας ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε πιο, να βελτιώσουμε τις πληροφορίες σε σχέση με τους καταναλωτές και να, γι' αυτό εισήγαγα την υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων Καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών. Ποια είναι η ιδέα πίσω από αυτό πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές, λέμε, οι πληροφορίες που θα πρέπει να είναι απλές, εύληπτες και αναγκαίες. Τίποτα το περιττό. Και να έχουμε εδώ, να αποφύγουμε περίπλοκες και περιτές πληροφορίες. Το πλαίσιο αυτό που θα δίνεται να είναι για τους καταναλωτές εύληπτο και να υπάρχει έτσι μια δυνατότητα προάσπισης των συμφερόντων τους και να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Δεύτερο, αυτό που έκανα είναι πρότεινα, πρότεινα μία η ιδέα αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης της ΣΕΠΑ, ώστε να είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε με εχέγγυα ότι όλοι όσοι θα εμπλέκονται στην αγορά και από πλευράς προσφοράς και από πλευράς ζήτησης να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να επηρεάζουν τη λήψη απόφασης, της αποφάσης. Και τέλος εισήγαγα ένα άρθρο που έχει ως στόχο τη δημιουργία κανόνων και κανονισμών τεχνικού χαρακτήρα που θα εκδίδονται από την ΕΒΑ ώστε να δημιουργηθεί ας το πω έτσι ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την λειτουργία αυτών των πληρωμών. Έτσι στόχος μου είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τρόποι να, να, να δημιουργηθούν προσκόμματα και εμπόδια σε όσους θέλουν να εισαχθούν στην αγορά και θα είναι νέο εισερχόμενοι στην αγορά και να υπάρχει μία μορφή, ένας τρόπος αναγνωρισμένος και ασφαλής για όλους να ε, δρουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο πληρωμών. Σε σχέση με τις αρχές λοιπόν, θεμελιώδεις αρχές που υιοθετούμε, δεν είναι μια κλειστή πρόταση αυτή, μια στεγανή πρόταση Είμαι απόλυτα ανοιχτό σε σχέση με επαφέ και φυσικά και με του σκιώδει εισηγητέ. Αυτή είναι η μέθοδο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μια ανοιχτή μέθοδο να ε, υποβληθούν, να κατατεθούν οι δικές τους προτάσεις, να υπάρξει μια αμφίδρομη δράση. Και τέλος τέλος θέλω να πω ότι σε σχέση με την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας που είναι μια περίπλοκη ευρύτερη οδηγία να μπορέσει να οδηγήσει σε μια ισορροπημένη σχέση, σε ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων. Να έχουμε από διαφορετικές θέσεις, ανταγωνιστικές θέσεις, αντίθετες απόψεις μεταξύ τους να οδηγηθούμε σε μια σύγκληση και μια συνένεση. Βασίζομαι στην υποστήριξη των σκιωδών εισηγητών και των συναδέλφων αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να το πετύχω αυτό. Σας ευχαριστούμε, Διέγο. Τώρα θα λάβουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές. Θα δώσω τον λόγο λοιπόν στους σοσιαλδημοκράτες πρώτα. σκιώδεις εισηγητές και μετά από πλευρά των ε, υπόλοιπων θα γίνουν οι παρεμβάσεις. Έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Ο κύριος Μπαντίνη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς ε, εσάς κύριε Σιγητά, για την ποιότητα της έκθεσής σας. Και χαιρετίζω και την όλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει ένα νομιόμορφο αποτελεσματικό ανταγωνιστικό σύστημα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθώ σε πολλά σημεία τα οποία προκαλούν μια κάποια ανησυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα όριο 0,3% ε, για τις πιστοτικές κάρτες και ένα ανώτατο όριο 0,2% για τις χρεωστικές κάρτες. Στα όρια όμως αυτά θα έπρεπε ουσιαστικά να έχουμε λάβει υπόψη μας διάφορους ε, οικονομικούς παράγοντες υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη. Εξελίσσονται διαφορετικά οι εθνικές αγορές, υπάρχουν διαφορετικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών και σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται διαφορετικά επιστοτικές κάρτες. Για παράδειγμα, στη Γερμανία το τέλος είναι 1,8%, στην Δανία 0,1%, στην Κροατία, τη χώρα μου, οι διατραπεζικές προμήθειες μπορούν να φτάσουν ακόμα και το 7%. Ποιες είναι οι συνέπειες λοιπόν όλων αυτών. Έχουμε ορισμένους εμπόρους οι οποίοι μπορούν να κάνουν ε, εκπτώσεις, προσφορές, ακόμα και τις τάξεις του 20% και παραπάνω, αν ο καταναλωτής αποφασίσει να πληρώσει μετρητά. Προτίμηση ουσιαστικά δίνεται Κυρίω τα μέτρητα ευνοείται αυτή η συναλλαγή και όχι η συναλλαγή με πιστοτικέ ή χρωστικέ κάρτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να αυξηθεί η ασφάλεια ή και ενημέρωση ή πρόσβαση σε πληροφορίε είναι ευπρόσδεκτη. Αποτελεί αυτό να το δικαίωμα των καταναλωτών. Δεν μιλάμε όμω μόνο για προσβασιμότητα, αλλά και για την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών. Θα πρέπει να αποσαφινιστούν οι κανόνε και θα πρέπει οι καταναλωτέ να είναι σε θέση να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές τις οποίες κάνουν. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ουσιαστικά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουμε τα αναμενόμενα ωφέλη. Θεωρώ ότι η οδηγία αυτή πάντω ευνοεί περισσότερο του εμπόρου και όχι τόσο του καταναλωτέ. και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε εμεί την όλη εργασία που κάνουμε εδώ πέρα του ίδιου καταναλωτέ. και α μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να μπορούν να γίνονται προσφορέ και να μειώνονται και οι τιμέ για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αν όμω, τα τέλη κυμαίνονται αυτή τη στιγμή από 0,2% σε 1,8% κάποιο καταβάλει τελικά το τίμημα. Ποιο θα καταβάλει το τίμημα αυτό, οι καταναλωτέ ή θα βρεθούν κάποια άλλοι εναλλακτικοί τρόποι για να μην επομιστούν το τίμημα αυτό οι καταναλωτέ. Το σημαντικό είναι μέσω τη πρωτοβουλία αυτή να προστατεύσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, του μικρομεσαίου εμπόρου, καθώ επίση και του καταναλωτέ. Η χρονική περίοδο των τεσσάρων ετών, καθώ επίση και η ρήτρα αναθεώρηση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τις ε, διατραπεζικές προμήθειες, η προβλεπόμενη χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να περιοριστεί. Ιδίω όσον αφορά τις διατάξεις εκείνες που έχουν να κάνουν με την προστασία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τελική απόφαση που θα λάβουμε θα είναι η κατάλληλη, η σωστή απόφαση και ότι θα αποφύγουμε τυχόν αρνητικές δυσμενείς επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τους μικρούς μεσαίους εμπόρους. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι στην ε, καθόλα καλή έκθεση που έχουμε μπροστά μας υπάρχει ένα κάποιο περιθώριο για περαιτέρω απλούστευση για να χρησιμοποιήσω την ορολογία που χρησιμοποιήσει ο κύριο Ζάλμπα. Θα πρέπει να απλουστευτεί περισσότερο το προτινόμενο λοιπόν κείμενο και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλτίνη. Ο εισηγητής εκ μέρους των σοσιαλιστών, ο κύριος Λούντβικστον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, καθώς επίσης και τον σκιώδη εισηγητή, τον κύριο Φέιο, για τις πολύ καλές προτάσεις που κάνανε θεωρώ ότι το κείμενο αυτό αποτελεί μια καταπληκτική εφετηρία για το μελλοντικό μα έργο. Ξέρω ότι δίστανται οι απόψει μα σε διάφορα σημεία, αλλά για πάρα πολλού τομεί νομίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν κάποιο συμβιβασμό. Πρώτη παρατήρηση γενική φύσεω. Επεξεργαζόμαστε την προτινόμενη λοιπόν αυτή νομοθεσία και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε και εδώ μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κατακαιρματισμό σε 28 διαφορετικές αγορές. Αυτό είναι πραγματικά παράλογο, περιορίζει τον ανταγωνισμό καθώς επίσης και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Προφανώς, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια πλήρως λειτουργούσα, απολύτως ενιαία αγορά, αλλά το καλό θα ήταν να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι σαφές για μένα. Περνάω τώρα στο πιο σημαντικό τμήμα της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε με τα τριμερή συστήματα και κυρίως με τους ε, τρίτους φορείς, τους TPPs. Οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα, σαν αυτό το οποίο θέλουμε να θεσπίσουμε, πρέπει να διέπεται από γενικούς κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν καλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπεται επαφή ανάμεσα στους παρόχους πληρωμών και τους TPPs, τους τρίτους φορείς. Ο εισηγητής ουσιαστικά κάνει θετικές προτάσεις προς αυτό, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν ανα πάσα στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο ίδιος ο καταναλωτή θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει πλήρως πω έχουν τα πράγματα και να προστατεύεται πλήρως από κάθε άποψη. Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ποιος ευθύνεται γιατί, σε περίπτωση που έχουμε μια παρατυπία ή μια συναλλαγή η οποία δεν θα εξελιχθεί θετικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόταση τη σχετική του ηγητή. Ένα άλλο σημαντικό σημείο έχει να κάνει με, τις, με τα επιπλέον τέλη. Δεν συμφωνώ εδώ με την πρόταση του εισηγητή. Πιστεύω ότι τα επιπρόσθετα αυτά τέλη δεν διδραματίζουν κανέναν θετικό ρόλο στην αγορά. και ούτε λειτουργούν ω λογικοί μηχανισμοί ελέγχου ή καθοδήγησης όπως λέγεται. Δημιουργούν απλώ περαιτέρω προβλήματα. Επομένω, τα τέλη αυτά συναλλαγή θα πρέπει να αποφευχθούν γιατί πολλέ φορέ απλώ τα χρησιμοποιούν οι φορεί πληρωμή, παροχή των υπηρεσιών αυτών πληρωμή για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα από τον ίδιο τον καταναλωτή. Θα πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν το ζήτημα αυτό ακόμα περισσότερο. Στα κράτη-μέλη εκείνα όπου οι κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει αυτά τα τέλη συναλλαγών είδαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Αν πραγματικά λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά πληρωμών, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα επιπρόσθετα τέλη συναλλαγών για ορισμένες κάρτες θα απαγορευτούν εντελώς. Και νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενό της. Ουσιαστικά θα πρέπει πραγματικά να απαγορεύσουμε τις επιπρόσθετες ε, προμήθειες και για όλες τις υπόλοιπες πληρωμές, όπως ακριβώς λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενό της. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, ευνοϊκές συνθήκες για το καταναλωτή δηλαδή, και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία ρύθμιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η απαγόρευση αυτή των επιπρόσθετων τελών όσον αφορά τις συναλλογές θα πρέπει να προβλέπεται για όλους τους ε, εμπόρους και να μην τους επιτρέπει ουσιαστικά να κάνουν μια κάποια επιλογή της μεθόδου εκείνης που θα τους αποφέρει περισσότερα χρήματα εις βάρος των καταναλωτών. Τώρα όσον αφορά τους ορισμούς, απουσιάζουν πολλοί ορισμοί και αυτό αποτελεί αδύναμο σημείο της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχαίρω τον εισηγητή, ο οποίος προσπάθησε να διορθώσει το πρόβλημα αυτό επεξεργαζόμενος κάποιους ε, ορισμούς νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο. Να καταφέρουμε να καταρτήσουμε κάποιους σωστούς ορισμούς. Οι προτινόμενοι ορισμοί, οι λίγοι προτινόμενοι ορισμοί νομίζω ότι δημιουργούν τελικά κάποια προβλήματα και ουσιαστικά υπερβαίνουν το στενόριο των ορισμών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο σαφές νομοθετικό πλαίσιο για το καταναλωτή. Όσον αφορά τώρα τις επιγραμμικές online συναλλαγές, πάλι πολύ καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαφώς χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, καλύτερη ενημέρωση, περισσότερη διαφάνεια. ακόμα και αν οι κανόνες δεν μπορούν να καλύπτουν πάντα και τις δύο πλευρές μιας συναλλαγής, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε αν μη τι άλλο στη μία πλευρά, προκειμένου στον καταναλωτή, να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Ο εισηγητής προσπάθησε μέσω των ε, προτάσεών του να μειώσει και το τέλος που επιβαρύνει τους καταναλωτές από 150 ευρώ σε 50 ευρώ σε περίπτωση παρατυπίας ή ε, απατηλής συναλλαγής. Αυτό είναι πολύ καλό και νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε και άλλους τρόπους συνεργασίας του καταναλωτή και του εμπόρου σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα απάτηση παρατυπιών. Χαίρομαι επίση πάρα πολύ που βλέπω ότι έχουμε καταργήσει πάρα πολλέ εξαιρέσει ή έχουμε μειώσει σε ορισμένε περιπτώσει τις διάφορε εξαιρέσει που ισχύανε σε προηγούμενες οδηγίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι περισσότεροι συναλλασσόμενοι εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και έχουμε σημειώσει και πρόεδρο όσον αφορά τα ATM, τις συσκευές ανάληψης χρημάτων. Προσβλέπω σε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες και συγχαίρω για άλλη μια φορά τον εισηγητή που δημιούργησε μια πολύ καλή αφετηρία, πολύ καλή βάση εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ βλέπω φίλους από την Αβάρα. Καλώς ήρθατε και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Η κυρία Χιλφέλτ έχει τώρα το λόγο που είναι σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρου των φιλελεύθερων και για τις δύο εκθέσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους εισηγητές για τις προτάσεις τους. Νομίζω ότι μένει πολλή δουλειά να γίνει και για τις δύο προτάσεις. Πρόκειται για ένα θέμα αρκετά τεχνικής φύσεως, αλλά είναι και πολιτικής φύσεως. Γι' αυτό και υπάρχουν διαφωνίες προς τα που θέλουμε να κατευθεθούμε. Μια γενική παρατήρηση είναι ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γενικά μιλώντας, έχουν καλή βάση, αλλά εδώ με δύο υποσημειώσεις. συζητάμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις αυτές, προσπαθούμε να βρούμε νέες μεθόδους πληρωμής, ενώ στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν τα bitcoins που μπορεί να εξαφανιστούν. Αλλά, πάση περιπτώσει, να μην ξεχνάμε ότι οι εξελίξεις πάνε πιο γρήγορα από ό,τι πάμε εμείς. Συνεπώς πρέπει να επιταχύνουμε το ρυθμό μας και να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις, να νομοθετούμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Όσον αφορά τις προτάσεις των εισηγητών τώρα. Για το εύρος εφαρμογής πρώτα απ' όλα. Η συζήτηση επικεντρώνεται από ό,τι φαίνεται κυρίως στο κατά πόσο τα τριμερή συστήματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ή όχι. Και ίσως και κάποια άλλα. Αναρωτιέμαι, μήπως μπορούμε να βρούμε μια διατύπωση όπου οποιοδήποτε σχήμα θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εφόσον φτάσει σε κάποιο όριο, το οποίο να καθορίζεται είτε από το μερίδιο στην αγορά, που βέβαια είναι δύσκολο να καθοριστεί, ή από τον όγκο, ή τέλο πάντων κάποιο μπορεί να έχει μια άλλη καλύτερη ιδέα. Διότι βλέπετε, θα ήθελα μια λύση που. Μάλλον δεν θα ήθελα μια λύση που να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα ή να τα αποκλείουμε όλα. Θα ήθελα μια διάμεση λύση. Δεύτερον, για το επίπεδο των διατραπεζικών προμηθειών. Δεν ξέρω ποιο είναι το καλό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι αυθαίρετο. Ακούσαμε τις εξηγήσεις της Επιτροπής για το πώς φτάσανε στο 0,2 και 0,3%, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι. Εγώ λέω ότι το επίπεδο θα πρέπει να είναι 0% εκτός εάν δικαιολογείται ένα άλλο ποσοστό. Ή ίσως να σκεφτούμε κάποιο σταθερό ποσοστό, τουλάχιστον για τις χρεωστικές κάρτες. Δεν ξέρω πάντως αν πρέπει να δεχτώ το 0,2 και 0,3% σαν κάτι που είναι έτσι και δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν με ενθουσιάζει η πρόταση για το μεσόρο. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι λύση και αν τελικά κρατήσουμε πρέπει να έχει κάποια αιτιολόγηση. Να φαίνεται γιατί καταλήγουμε σε αυτήν και όχι σε άλλη. Ο εισηγητής προτείνει να διαγράψουμε κάποια σημεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Εμένα αυτό μου δημιουργεί απορία, γιατί όλοι συμφωνήσαμε, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά και να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αποκλήσεις. Οπότε δεν βλέπω γιατί εσείς θέλετε να διαγραφεί αυτό. Έπειτα μια παρατήρηση που ισχύει και για τις δύο εκθέσεις. βρίσκω ότι εδώ δίνουμε ε, δεσπόζουσα θέση στις τράπεζες. Γι' αυτό άκουσα προσεκτικά την πρόταση του κυρίου Φέια για τη ΣΕΠΑ, για τον νέο χώρο πληρωμών σε ευρώ. Είναι επιχειρήσεις. Έτσι κι αλλιώς. Συνεπώ, να έχουν μεν κάποια θέση, αλλά όχι δεσπόζουσα. Και τώρα γρήγορα για τις προτάσεις σας όσον αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες. Εγώ είμαι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νομική αποδέσμευση. Προτείνω την πρόταση της Επιτροπής επίσης όσον αφορά το co-badging. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο ξεκάθαρο το πώς θα λειτουργήσει το θέμα τελών για τις κάρτες. Γιατί κάποιοι λένε ότι αν αλλάξει ο κανόνας προς μία κατεύθυνση δημιουργείται μεγαλύτερη σύγχυση. Ναι, αλλά και προς την άλλη κατεύθυνση αν κάνετε μια αλλαγή πάλι προκαλείται σύγχυση. Οπότε εγώ θέλω να ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση για όλους. Για το PSD συμφωνώ με τόσα είπαν οι προλαλήσαντες για το εύρος εφαρμογής που νομίζω ότι πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ευρύ το εύρος της οδηγίας αυτής για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Εναρμόνιση των ε, τελών θα ήμουν υπέρ μιας γενικής απαγόρευσης και όχι τα κράτη-μέλη να έχουν την ελευθερία να το καθορίζουν αυτό γιατί τότε παραμένει η κατάσταση που ισχύει και τώρα, κάτι που δεν θέλουμε. Πρόσβαση στις πληροφορίες των λογαριασμών πληρωμής. Εδώ ας ακούσουμε τον επόπτη προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει κάποιες πρακτικές προτάσεις Η Επιτροπή μας μάλιστα νομίζω ότι θα έπρεπε να ζητάει την άποψη του επόπτη αυτού πολύ πιο συχνά από ό,τι το κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Το θέμα της ευθύνης αυτό επίσης θα ήθελα να το δούμε περισσότερο. Δεν είμαι πεπισμένη ότι είναι καλές οι προτάσεις που γίνονται ώστε το κύριο βάρος της ευθύνης να είναι στους παρόχους και όχι στις τράπεζες. Τα άλλα τάπα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Σοφή. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, ο κύριος Γκυγόλ, σωστά. Ευχαριστώ. Κάπως αμήχανα αισθάνομαι εξ ονόματος PSD2 Jean Paul Bechet, δεν βάζω τον λόγο και προσπαθώ να ομολογήσω ότι για τις, ε, τις ρυθμίσεις ε, των μετακυλιόμενων ή εισπρατώμενων τελών ε, θα ήθελα να παρέμβω. Δεν είναι οι δικές μου απόψεις, είναι οι απόψεις συναδέλφων. Πρώτα για την οδηγία για τις πληρωμές αυτές συμφωνούμε ότι με τον εισηγητή ότι είναι πολύ κατακαιρματισμένη ακόμα η αγορά αυτή για τους καταναλωτές και πάρα πολύ επικεντρωμένη από την άλλη πλευρά ε, ε, στις επιχειρήσεις σε σχέση με τους καταναλωτές δεν αποβαίνουν ωφέλη και σε σχέση με τις υπηρεσίες ε, και την ε, μετάθεση πληρωμών ε, θα πρέπει εδώ να δούμε εναλλακτικέ δυνατότητες για μειωμένα τέλη. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες σε κάποια κράτη-μέλη και είναι ασφαλής και υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευράς καταναλωτών. Πρέπει όμως να ρυθμιστούν με τον πιο σωστό τρόπο και να επανενταθούν σε ένα ευρωπαϊκό ενιαίο πλαίσιο. Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών πρέπει να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια. Ποιος θα υπεύθυνο για ποιο πράγμα. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια πληρωμών, την ε, ε, λογοδοσία, την ε, υπευθυνότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για το εύρο, για το φάσμα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί αυτό στην πρόταση και είναι κύριος στόχος να μεριμνήσουμε ότι θα γίνει αυτό από πλευρά μα Για το άρθρο 3 και το θέμα του αρνητικού ε, εύρους, γενικά εγκρίνουμε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να υπάρξει ε, ένα, μια μείωση του φάσματος αυτού. Δεν κατανοούμε γιατί θέλει ο εισηγητής να διαγραφεί το εδάφιο για την χρέωση όσον αφορά αυτά τα τέλη και όσον αφορά και το εδάφιο 13 Επίσης συμφωνούμε με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαναδιοριστεί η εξαίρεση για τις τηλεπικοινωνίες στο άρθρο 3 αλλά πιστεύουμε ότι η έννοια των επικουρικών υπηρεσιών, auxiliary services, δεν επαρκεί σε σχέση με, για παράδειγμα, τα ποσά που προτείνονται 50 ή 200 ευρώ που πρέπει να δικαιολογούνται. Μπορεί να εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω και να δώσει διευκρινήσεις Τώρα, σε σχέση με τα δικαιώματα των ε, ε, καταναλωτών που πρέπει να τους ε, παρέχονται αγαθά ή υπηρεσίες και που δεν μπορούν να, να ανταλλάσσονται σε σχέση με μετρητά για το άρθρο 3, το εδάφιο K. Αυτό που υπάρχει στη Γαλλία, τίτλο service, τίτλος υπηρεσίας, φαίνεται ότι εξυπηρετεί την ε, ε, η παροχή υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να θέσουμε κάποια ε, ερωτηματικά όσον αφορά την εξαίρεση για την χρήση travelers checks, δηλαδή επιταγών, ταξιδιωτικών επιταγών. Επίσης έχουμε και ερωτήματα όσον αφορά το εδάφιο 37 από τις, το κείμενο του εισηγητή πράγμα το οποίο θα ήταν οπισθοδρόμηση αν εγκρινόταν. Τον ορισμό, τους ορισμούς στο άρθρο 4 στη συνέχεια, για αυτούς τους ορισμούς εμείς θέτουμε ερωτήματα όσον αφορά ευαίσθητα στοιχεία πληρωμών δεν έχω ξαναδεί τέτοια πιο περίεργη ε, διατύπωση για το και από πού θα ε, προερχόταν κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τον επόπτη προστασίας προσωπικών δεδομένων για την λειτουργία με μια τέτοια πρόταση, θεωρούμε ότι αυτό θέτει προβλήματα και είναι ένα πραγματικά προβληματικό ε, κείμενο. Όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση, τη διαχείριση, το άρθρο 94α και το αντίστοιχο, την, η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση σε σχέση με τα τέλη και τον ανταγωνισμό σήμερα. Υπάρχει νομίζω περιθώριο να υπάρξει συμφωνία με τον εισηγητή όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη 5 και το 74α στοχεύει ο εισηγητής να, να διασφαλιστεί ένας ενεργός ρόλος όσων εμπλέκονται ε, σε σχέση με τον φορέα αυτό. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι υπήρξαν υποσχέσεις που δόθηκαν σε σχέση με την νομοθετική διαδικασία ρύθμισης ε, του ΣΕΠΑ. Θα το θυμάσαι και εσύ Σοφή πόσο κράτησαν αυτές οι μακρές διαπραγματεύσεις. Έδωσε και μια δήλωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να ξέρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού βρίσκεται, πώς τοποθετείται και ποιες είναι οι προοπτικές αυτής της ε, δράσης της. Ε, μας είχαν δοθεί υποσχέσεις ε, και όταν βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν και νέα στοιχεία όσον αφορά την ε, ε, σύνθεση ε, των τελών, θα θέλαμε να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Σε σχέση με το 7α και το 94β θα πρέπει να πληροφορούνται καλύτερα για τα δικαιώματά τους οι καταναλωτές και πρέπει να αναπτυχθούν τα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα και αν δεν θεωρούμε ότι ο όρος φυλάδιο, leaflet, είναι εκείνο το οποίο είναι το πιο ενδεδειγμένο σε αυτό το πλαίσιο και ηλεκτρονικά μέσα επίσης θα μπορούσαν ε, να ήταν ε, ενδεδειγμένα. Δεν κατανοούμε γιατί ο εισηγητής θέλει να διαγράψει την αναφορά σε ρυθμίσεις προστασίας των καταναλωτών στο σημερινό ενισχύ νομικό πλαίσιο σε σχέση με την αιτιολογική σχέση, ε, σκέψη 42. Μετά σε σχέση με το άρθρο 26 και το 63 έχουμε εδώ μια κλασική περίπτωση ε, αντίφαση, αντίφασης. Θεωρούμε ότι οι εθνικές υπηρεσίες προστασίας καταναλωτών πρέπει να έχουν δικαιώματα και ε, αρμοδιότητες άμεσα να ενεργοποιούνται εκεί όπου δεν υπάρχει δυνατό, δεν εφαρμόζεται το PSP. Ε, ναι, είναι πραγματικά πρέπει να πω αξιοπερίεργη αυτή η κατάσταση. Μετά για το άρθρο 34, το βάρος της απόδειξης για τις απαιτήσει πληροφόρησης, ενημέρωσης το βάρος αυτό δεν μπορεί να από πλευρά των κρατών μελών να απομένει στην PSP όπως προβλέπεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι εθελοντική η εφαρμογή αυτών. Αν θέλουμε μια πραγματικά ενιαία εσωτερική αγορά για τις πληρωμές, ας υπάρχουν ενιαίοι κανονισμοί σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τους καταναλωτές. Μετά για τα τέλη στο άρθρο 94β, αιτιολογική σκέψη 28α. Εδώ τίθενται, δημιουργούνται κάποια πρόσθετα κόστη. Ενώ δεν είμαστε κατά της ε, βασικής ε, αρχικής πρότασης, θεωρούμε ότι ε, οι καταναλωτές θα πρέπει να εντάσσονται στην ομάδα εργασίας EBA και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επιπτώσεις προτύπων επιχειρήσεων και μετά η επιστροφή για συναλλαγές που ξεκινούν σε σχέση με το άρθρο για παράδειγμα 67 και όσα προβλέπει. Παρότι με την πρόθεση των προτάσεων της Επιτροπής συμφωνούμε, θα πρέπει να κλείσουν οι πόρτες και παράθυρα χωρίς να δίνουμε, δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε απεριοριστά δικαιώματα. Ε, για, το επόμενο άρθρο δεν κατανοούμε την πρόθεση του εισηγητή να επιτρέπεται στις CNAs να περιορίζονται οι απαιτήσει για πληρωμές υπηρεσιών σε σχέση με την υπέρβαση ενός κατοφλίου 600 ευρώ στο άρθρο 9 αυτό. Ίσως θα μπορούσατε να επεξηγήσετε περαιτέρω αυτό την λογική που εμπνέει εσάς να καθορίσετε αυτό το κατόφλι. Μετά η πρόσβαση σε τέτοιου είδους συστήματα πληρωμών. Μία από τις τροπολογίες του εισηγητή έχουμε την εντύπωση ότι κάποιες τροπολογίες ε, εμπνέονται από τις ε, ε, καταχρήσεις ή υπερβολές στην αγορά. Δεν θεωρούμε ότι είναι το πιο σκόπιμο να υπάρχουν τέτοιου είδους διατάξεις. Θα θέλαμε να έχουμε ένα ισοδίκαιο πλαίσιο ε, δραστηριοποίησης όπως οι διατάξεις ε, για τις πιστοτικές κάρτες ε, με ευανάγνωστο τρόπο ανάγνωσης του, του, IBAN και των σχετικών για, τα, για τους λογαριασμούς στοιχείων. Για το επόμενο άρθρο πραγματικά έχουμε πρόβλημα με τη, όσα κινούν τον εισηγητή να προτείνει αυτό. Τώρα για τον έλεγχο IBAN δεν είναι εμπιστευτική αυτή η πληροφορία σε κάποια κράτη-μέλη. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, ερωτήματα όσον αφορά την ε, λογοδοσία, την υπευθυνότητα και για την καινοτομία στο άρθρο 58. Η πράσινοι πάντα ήταν υπέρ ανοιχτών πρωτοκόλων, όπως το Linux, Linux για παράδειγμα. Linux. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή ότι οι διαδικασίες πρέπει να καθορίζονται από τα PSPs οι τεχνολογικές διατάξεις πρέπει να μπορούν να συνδιαμορφώνονται και από ενδυνάμει ανταγωνιστές μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Το τέλος όσον αφορά τον κανονισμό για τα τέλη τα οποία θα εισπράττονται. Περνάω στον κανονισμό τώρα. Το 0,2% για την χρέωση, για την ε, δημιουργία του κόστους αυτού που προκαλείται στη Γερμανία και είναι υψηλότερο Έχουμε κράτη-μέλη με συστήματα που λειτουργούν καλό σήμερα. Θα έπρεπε να αποσαφινιστεί ρητά και κατηγορηματικά ότι επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να θέσουν χαμηλότερα ε, κατόφλια, χαμηλότερα επίπεδα τελών. Υπάρχουν, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος από την Κροατία, χώρες όπου υπάρχουν τέτοιες ε, χαμηλότερες χρεώσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης ε, της ίσπραξης, ε, των διατάξεων ίσπραξης αυτών των τελών ή να καθοριστούν και χαμηλότερα ποσοστά ίσπραξης. Αυτό θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη αποδοχή από τις επιχειρήσεις ε, της ε, χρήσης αυτών των καρτών και θα διευρύνει τις δυνατότητες για τους καταναλωτές. Η πρόταση για ένα σταθμισμένο μέσο όρο είναι ενδιαφέρουσα, αλλά απομένει να δούμε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ποιος θα καθορίζει τον επιμερισμό τελών σε σχέση με ε, διάφορες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όσον αφορά το co budgeting στο άρθρο 8. co budgeting σημαίνει συνδυασμό διαφορετικών, ε, ε της πληρωμής διαφορετικών ε, ε, λογοτύπων. Για παράδειγμα, Cash και Maestro για τη Γερμανία. Έχει ισχυρά επιχειρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλιστεί η λειτουργία του co-budgeting. Είναι μία από τις δυνατότητες ώστε να διασφαλιστεί ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Τώρα, για το, την ανησυχία να διαγραφεί αυτή η πρόταση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την πιο αποτελεσματική διαδικασία ε, πληρωμής. Η διαγραφή θα μπορούσε να απαγορεύσει σε νεοεισερχόμενους να εντάσσονται σε μια τέτοια κάρτα. Αυτό θα δυσχέρενε την πρόσβαση στην αγορά για νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Και μετά σε σχέση με την ε, χρήση αυτών των καρτών υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ και πάλι προτείνει ο εισηγητής να διαγραφεί αυτό το εδάφιο. Η επεξήγηση είναι ότι θα απολεστεί η εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο αν δεν γίνονται δεκτές οι κάρτες των καταναλωτών. Αυτό τι σημαίνει όμως σημαίνει ουσιαστικά να υποχωρήσουμε σε σχέση με την κατάχρηση της αγοράς ε, κάποιων επιχειρήσεων και δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέλη, τέτοιου είδους ε, καταχρήσεις στα τέλη οι καταναλωτές. Αν πιστεύει πραγματικά ο εισηγητής στον ανταγωνισμό, προγράμματα καρτών με τόσο αδικαιολόγητα υψηλά τέλη, δεν είναι σωστή η διατύπωση αυτή από πλευράς ε, ε, συντακτικής, συντάξεως και σε σχέση λοιπόν με την μη ευρύτερη αποδοχή αυτών των καρτών λόγω των υψηλότερων αυτών τελών είναι σαφές τώρα το νόημα αυτής της πρότασης. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη θετική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρου του ECR. Ο κύριος Άσλι Φόξ. Η κυρία Άσλι Φόξ. Ευχαριστώ. Όχι, η Άσλι Φόξ είναι στην ΕΜΚΟΠ. Ο κύριο Άσλι Φόξ είναι στην ΙΜΚΟ, εγώ τον αντικαθιστώ. Το ΕΣΥΑΡ λοιπόν ανησυχεί για τον κατακαιρματισμό της αγοράς αυτής με τα εθνικά σύνορα ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες, κάτι το οποίο πλήττει τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Εμείς στηρίζουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστούμε τον εισηγητή για το έργο του. Γιατί εμεί ακούμε τις ε, απόψεις και διαμορφώνουμε την άποψή μας. Ο Άσλε ανησυχεί για το γεγονός ότι οι τραπεζικές προμήθειες δεν μπορούν να προστατεύσουν ε, τον ε, ανταγωνισμό και είναι πολύ σκεπτικιστής όσον αφορά τα θετικά από τη χρήση, την χρήση των κρατών. Αν πάντως καταλήξουμε κάπου, μας ενδιαφέρει να μην υπάρχουν ε, αρνητικές συνέπειες και αυτό μπορεί να γίνει αν είναι χαμηλό το ποσοστό 0,3%. Τονίζει ότι οι πιστοτικές κάρτες δεν είναι ρευστό και δεν θα πρέπει να συγκρίνουμε το κόστος μεταξύ των ε, δύο. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι με το ποιον τρόπο πληρώνονται οι πιστοτικές κάρτες και συμφωνεί και με τους συναδέρφους για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρέπει να δικαιολογήσει τα ποσοστά που προτείνει και θα ήθελε περισσότερες αποδείξεις. Γιατί αυτά τα ποσοστά δηλαδή και όχι άλλα. άλλα θέματα, το ECR θεωρεί ότι το διασυνορικό ζήτημα πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα με το ωφέλη και το κόστος, όπως επίσης να δούμε το θέμα του ανταγωνισμού στις διάφορες εθνικές αγορές, γιατί υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει υπερβολική πίεση στις χώρες μέλη. Σχολιάζει ότι η προσέγγιση του εισηγητή όσον αφορά το co-badging είναι πολύ θαραλέα ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που εκφράζουν και καλώ τις εκφράζουν όλες οι πλευρές. Τώρα για την έκθεση ΦΕΙΟ. Ευχαριστούμε για την εκτενή δουλειά σας με όλες αυτές τις τροπολογίες. Προσβλέπουμε στην οδηγία αυτή προκειμένου να υπάρξουν οι ίδιες, ε, να ισχύουν τα ίδια για όλες τις πλευρές και μπορούμε να στηρίξουμε πολλές από τις τροπολογίες όσον αφορά το νομικό καθεστώς των παρόχων πληρωμών, τα τρίτα μέρη, το θέμα επίσης της ευθύνης των TTP, να υπάρχει ευθύνη απέναντι στους πελάτες εφόσον γίνει μια πληρωμή που δεν επιτρέπεται κανονικά. Βέβαια παραμένουν θέματα για τις συμβατικές ρυθμίσεις ανάμεσα στα TTP και τους παρόχους. Ο εισηγητής και οι σκιώδης πιστεύω ότι θα το συζητήσετε πολύ καλά αυτό. Τέλος, ο Άσλε σημειώνει ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη η οδηγία PSD 2 θα διευκολύνει τους, θα προσφέρει διευκόλυνση στους κατανοητέ πολύ περισσότερο από ό,τι περιεχόμενο για δωρές που γίνονται με ένα κείμενο κάτι το οποίο διευκολύνεται και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη χώρα μου και φαντάζομαι όχι μόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι δικτύων θα εμπίπτουν σε ρυθμίσεις και από πλευράς οικονομικών υπηρεσιών και από πλευράς Telecom. Και οι συναλλαγές πρέπει να είναι, όταν πρόκειται για δωρές, πολύ χαμηλό το κόστος πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις αυτού, όταν δηλαδή πρόκειται για φιλανθρωπικές δωρές. Ο Άσλη θα ήθελε να αντιμετωπίσει και αυτό το θέμα ο κύριος στην πρώτη του έκθεση. Ελπίζει ότι οι συνάδελφοι θα δεχτούν τροπολογίες του προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οπότε η FD τώρα. Ο κύριος Ντέχο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σκιώδεις, αγαπητέ κύριε Σιγητά και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχα πει ότι θέλω να κρατήσω ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και θέλω να πετύχω μια βελτίωση του ανταγωνισμού ώστε οι καταναλωτές να έχουν καλύτερη επιλογή όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών. Σήμερα όμως θα επικεντρωθώ στην πρόταση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών. Καταλαβαίνω σε κάποιο βαθμό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ρυθμίσει αυτές τις συναλλαγές με τη χρήση καρτών, τις διασνοριακές, αλλά δεν είμαι πεπισμένος ακόμα ότι πρέπει πραγματικά σε εθνικό επίπεδο να θέσουμε όρια όσον αφορά τις εγχώριες πληρωμές με χρήση καρτών. Οι εθνικές αυτές προμήθειες δεν αποτελούν δική μας αρμοδιότητα σε καμία περίπτωση. Αν όμως τελικά εγκρίνουμε μία νομοθεσία κοινοτική και για τις εθνικές προμήθειες, τότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές αγορές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει τελικά το κράτος μέλος να έχει τον τελευταίο λόγο, εφόσον αυτό έχει την απόλυτη αρμοδιότητα. Ας δούμε επίσης και τα διαφορετικά επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει πάλι ένα κίνδυνο αναστάτωση του επιχειρηματικού μοντέλου. Κάποιο πάντα θα πρέπει να καταβάλει ένα τίμημα για την παροχή μια υπηρεσία και αν αρμονίσουμε τι προμήθειε θα πρέπει μη τι άλλο να αποφύγουμε την αύξηση του κόστου για τον καταναλωτή. Παράλληλα όμω θα πρέπει να δώσουμε και σε επιχειρήσει, να διατηρήσουμε μάλλον το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο. Συμφωνώ με το σχέδιο έκθεσης όταν ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, όπου θα πρέπει να αξιολογείται και η επίπτωση στους καταναλωτές αλλά και στους εμπόρους. Ας μην ξεχνάμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων αυτών κάθε φορά που εμείς εγκρίνουμε μια νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα το co-badging, Σίγουρα τα όσα προβλέπονται είναι θετικά, αλλά θα πρέπει να έχουν θελούσιο χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τώρα τι κάρτε πληρωμών και το διαχωρισμό με του φορεί επεξεργασία, συμφωνώ εδώ πέρα με τον εισηγητή. Τέλο, στα πλαίσια τη νομοθεσία αυτή νομίζω θα δημιουργήσουμε πολλέ επιπτώσει στου καταναλωτέ και στον τρόπο που χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε πληρωμών. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν επεξεργαζόμαστε το ζήτημα αυτό, δεν θα πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Γι' αυτό σα ζητώ να παραταθεί η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών. Έχουμε ελάχιστε μέρε πριν τι χριστουγεννιάτικες διακοπέ για να καταθέσουμε τροπολογίε. Θεωρώ ότι δεν αρκεί ο χρόνος αυτός, επομένως αν γίνει να μα δώσει μια μικρή παράταση αυτό θα μα βοηθούσε όλου ιδιαίτερω. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σέμπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα πάρει το λόγο. Θέλετε το λόγο, έτσι δεν είναι. Ε, ένας από τους δυο σας, εσωτερική αγορά, ανταγωνισμός, όποια γενική διεύθυνση θα μιλήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω πρώτη εγώ το λόγο και θα μιλήσω εξ ονόματο τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τον Κανονισμό και ο συνάδελφό μου στη συνέχεια θα σα μιλήσει για την πρόταση οδηγία υπηρεσιών πληρωμών. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την έκθεση αυτή, την πολύ καλή συζήτηση την οποία είχαμε και τις δυνατότητες που μας δίνετε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις για την πρόταση. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε μια πρόταση κανονισμού εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι τραπεζικέ προμήθειε. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε όλα τα κρυφά τέλη τα οποία υπάρχουν. Πολλέ φορέ, ω καταναλωτέ, θεωρούμε ότι χρησιμοποιούμε εντελώ δωρεάν μια κάρτα πληρωμή και ότι αποφελούμαστε πλήρω των ωφελημάτων που επιφέρει η κάρτα αυτή. Στην πραγματικότητα όμως ο πολιτής ουσιαστικά πληρώνει μία προμήθεια σε μία τράπεζα και το ποσό της προμήθειας αυτής που πληρώνεται προς την τράπεζα διαφέρει πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε μια κάρτα Bangkok στο Βέλγιο, ο πολιτής θα πληρώσει μόνο 5 λεπτά. Αν πληρώσουμε όμως με μια American Express, τότε η προμήθεια αυτή μπορεί να φτάσει στα 2,5 ή ακόμα και τα 3 ευρώ για ένα ποσό 100 ευρώ και έχετε μια τεράστια ψαλίδα εντωμεταξύ πολλών διαφορετικών ποσών, προμηθειών που πρέπει να πληρωθούν για τη Visa, για τη Mastercard, για χρεωστικέ κάρτε, για ε, πιστοτικές κάρτε και το καθεξής. Έτσι λοιπόν τόσο εμπόρο, όσο και καταναλωτή το βάρος, μάλλον η προσπάθεια, η διεργασία είναι ακριβώς η ίδια. Χρησιμοποιείται απλώς μία κάρτα, αλλά τελικά ο έμπορος καταλήγει να πληρώνει μία προμήθεια που είναι εντελώς διαφορετική ως προς την κάρτα και ως προς το κράτος μέλος. Στο Βέλγιο γενικά οι προμήθειες είναι χαμηλές, αλλά στην Πολωνία ή στην Ουγγαρία μπορεί να είναι δεκαπλάσια τα τέλη τα οποία πρέπει να πληρωθούν από τον έμπορο, το λένε πολιτή εμείς προσπαθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβουμε τις διαφορές αυτές, να αναλύσουμε τις διαφορές αυτές. Για ποιο λόγο οι εμπορικές κάρτες είναι τόσο ακριβές, για ποιο λόγο οι χρεωστικές κάρτες δεν μπορούν να γίνουν λίγο πιο φτηνές, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να μειώσουμε τις ε, διατραπεζικές προμήθειες και ουδέποτε μας δόθηκε μια ξεκάθαρη εξήγηση για όλες αυτές τις διαφορές μεταξύ καρτών και μεταξύ χωρών. Αυτή είναι η κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα στην Ευρώπη. Τώρα, οι έμποροι, οι ελληνοπολιτέ που αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή έχουν και μια ακόμα δυσκολία. Πρέπει να πληρώσουν όλα αυτά τα τέλη, πρέπει να καταβάλουν όλε αυτέ τι προμήθειε και καταλαβαίνετε ότι αν το κατάστημά του είναι σε μια χώρα με ψηλέ προμήθειε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν όπω καταναλωτέ στην εσωτερική αγορά και να πάνε να ψωνίσουν σε μια άλλη χώρα. Δεν μπορούν να εγκαταστήσουν το μαγαζί του σε μια άλλη χώρα. γιατί ακόμα και να γίνει κάτι τέτοιο, ακόμα και να εγκαταστήσουν τελικά το κατάστημά του σε μια άλλη χώρα, πάλι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να καταβάλουν τις προμήθειε προβλέποντα στη χώρα προελευσής τους. Και αυτό λειτουργεί ιδιαίτερα αρνητικά για τους εμπόρους και ιδίω για τους νέου ερχόμενου στην αγορά. τι νέε δηλαδή κάρτε, τι νέε υπηρεσίε πληρωμών που θέλουν να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και που πρέπει πάλι να αρχίσουν να πληρώνουν τα τέλη τα οποία προβλέπονται στη χώρα τους. Αυτό ισχύει και για τις κάρτες, αλλά και για τις πληρωμές μέσω τηλεπικοινωνιών, αλλά και για τις online πληρωμές, μέσω διαδικτύου δηλαδή. Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει είναι ότι όχι μόνο έχουμε προβλήματα ανταγωνισμού, αλλά και προβλήματα προστασίας του καταναλωτή. Στην αρχή είπα ότι εμείς οι καταναλωτές θεωρούμε ότι όλες αυτές οι συναλλαγές είναι δωρεάν. Στην πράξη σας απέδειξα ότι δεν είναι. Μέσω της καταβολής των προμηθειών αυτών από τους εμπόρους πληρώνουμε και εμείς σαν καταναλωτές γιατί αναγκαστικά αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων που αγοράζουμε. Ξέρετε ότι ε, αν ο λιανοπολιτής, ο έμπορος πρέπει να πληρώσει μια προμήθεια επειδή εμείς χρησιμοποιούμε μια κάρτα, τότε αναλογικά θα αυξήσει τελικά και τις τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζουμε. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποιες πιο φτηνές κάρτες που πληρώνουν με μετρητά, τελικά χρηματοδοτούν αυτούς οι οποίοι πληρώνουν με μια πιο ακριβή κάρτα που χρησιμοποιούν μια χρυσή κάρτα, μια American Express και ούτε καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν το, το σύστημα αυτό προκειμένου να πιέσουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις πιο ακριβές κάρτες, αυτές που αποφέρουν δηλαδή στις τράπεζες πιο ακριβές προμήθειες, πιο υψηλές προμήθειες. Εμείς προσπαθούμε να ελέγξουμε τις προμήθειες αυτές και να ελέγξουμε τη χρήση των πιστοτικών καρτών, γιατί όπως σας είπα πολλές φορές μέσω της, χρή... χρήσης των καρτών αυτών, ορισμένοι πιο φτωχοί καταναλωτές πληρώνουν για τους πιο πλούσιους καταναλωτές, για τη χρήση των πιο ακριβών καρτών. Αυτά όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο της πρότασης. Να σας πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα δυσέλιδο φυλάδιο ακριβώς επειδή η όλη αγορά εδώ είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και υπάρχουν πολλές παραπλανητικές πληροφορίες, ένα υψηλό ποσοστό παραπληροφόρησης το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή στους καταναλωτές, όπου θέλουμε πάλι να αποφύγουμε ότι οι πιο φτωχοί καταναλωτές πληρώνουν τελικά το τίμα για τη χρήση των πιο πολύπλοκων ακριβών καρτών. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διανύμουμε περισσότερο το φυλάδιο αυτό προκειμένου να ενημερώσουμε καταλήλω τους ε, καταναλωτές. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, ας περάσω πραγματικά τώρα στι διατάξει και τις προτάσεις για την τροποποίηση του κανονισμού. Όσον αφορά τι προτάσει που γίνονται στην έκθεση, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο ο εισηγητή θέλει να διορθώσει κάποια πράγματα, να τροποποιήσει κάποιε διατάξει. Θεωρούμε πάντω ότι υπάρχουν κάποιε σημαντικέ ε, διατάξει οι οποίες ενδεχομένως να μην ε, επιφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ξέρετε ότι ε, μέσω κάποιων προσφυγών που έχουν γίνει για δύο σημαντικά παγκόσμια συστήματα πληρωμής έχουμε πλέον μια νομολογία η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί στα πλαίσια του κανονισμού. Αν όμως ε, υποβάλλουμε διατάξεις διαφορετικές, τότε ουσιαστικά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την ομολογία αυτή. Ουσιαστικά ο κανονισμός αυτός δεν θα προσθέσει τίποτα περαιτέρω από αυτά τα οποία προβλέπονται στο υφιστάμενο σύστημα, από όσα έχουν προκύψει μέσω των προσφυγών αυτών που έχουν γίνει. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα ήταν θετικό, γιατί έχουμε εντοπίσει πολλά προβλήματα, στα οποία τελικά δεν θα δινόταν μια λύση. Τώρα, ας περάσω σε όλα αυτά τα σημεία της πρότασης ένα προς ένα. Πρώτον, ορισμός για τις διασυνοριακές πληρωμές και αγορές. Αν αλλάξει τελικά όπως προτείνετε εσείς ο ορισμός αυτός, τότε ουσιαστικά θα αναφερόμαστε μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν την κάρτα τους σε μια άλλη χώρα. Επομένως ο ορισμός δεν θα καλύπτει την περίπτωση εκείνη όπου ένας έμπορος πηγαίνει στο εξωτερικό και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της τραπεζικές μεσάλης χώρας. Και αυτό είναι πρόβλημα γιατί ουσιαστικά διονύζεται μια κατάσταση όπου οι έμποροι δεν μπορούν να αποφεληθούν από την εσωτερική αγορά. Και αν η εξήγηση που δίνεται είναι ότι δεν θέλετε εσείς να επηρεαστεί αρνητικά η αγορά, τότε μάλλον δεν έχετε καταλάβει κάτι καλά. Γιατί εμείς θέλουμε να επηρεαστούν από τον κανονισμό αυτό οι αγορές. Θέλουμε ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά όπου θα αποφελούνται όχι μόνο καταναλωτές, αλλά και έμποροι και λιανοπολιτές όταν πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα, όταν εγκαθίστανται σε μια άλλη χώρα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, τα απόλυτα όρια τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προμήθειες θα πρέπει να μειωθούν στο 0,2% και το 0,3%. Λέμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα απόλυτο ανώτατο όριο. Η έκθεσή σας λέει να χρησιμοποιηθεί ανταυτού ένα σταθμισμένος μέσος όρος. Καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το προτείνεται αυτό. Γιατί στην, ένα σταθμισμένο μέσο όρο χρησιμοποιούμε και στη σχετική νομοθεσία για τον ανταγωνισμό στον τομέα αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επιτρέπουμε ακόμα μια ευελιξία. Υψηλότερε προμήθειε σε κάποιε περιπτώσει, χαμηλότερε προμήθειε σε κάποιε άλλε. Εν προκειμένου δεν ξέρω πώ θα λειτουργήσει όμω το, το, το σύστημα αυτό τη ευελιξία. γιατί ξέρετε ότι εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένε εταιρείε συμβούλων, οι οποίε προσπαθούν να κάνουν μία ανάλυση και να δουν τελικά ποιε προμήθειες χρησιμοποιούνται. Ξέρετε ότι για τον κανονισμό αυτό γιατί δεν μιλάμε για οδηγία, μιλάμε για καονισμό. θα πρέπει οι εθνικέ αρχές να λάβουν το ρόλο αυτό και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα περιέπλεκε πάρα πολύ το έργο των κρατών μελών. Επίσης, πώς θα καθορίσουμε το σταθμισμένο αυτό μέσο όρο, ανατομέα, ανακλάδο, για παράδειγμα, στα προκυπευτικά θα είχαμε διαφορετικό σταθμισμένο όρο από ότι στα αυτοκίνητα θα γινόταν ανασύστημα, ανακράτο μέλο. Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Θα ήταν καλύτερο για αυτό το λόγο να κρατήσουμε το σύστημα που εμεί προβλέπουμε, δηλαδή τα ανώτατα όρια. Τώρα, αν κάποιες τράπεζες συναντήσουν προβλήματα από το προβλεπόμενο αυτό σύστημα, τότε τα προβλήματα αυτά μπορούν να διορθωθούν μέσω των συγκεκριμένων αυτών απολύτων ορίων. Από πάρα πολλές απόψεις θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό είναι καλύτερο από αυτό το οποίο προτείνεται. Τώρα, όσον αφορά τον κανόνα Honor All Cards, ο κανόνας για την υποχρεωτική αποδοχή όλων των καρτών. Πολύ φοβάμαι ότι ε, η δική σας ε, η πρόταση τελικά δεν θα επιτρέπει στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν όλες τις κάρτες. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να αποφύγουμε είναι τελικά οι πιο φτωχοί καταναλωτές να καταβάλουν το τίμημα για τις πιο ακριβές κάρτες, αυτές δηλαδή οι οποίες περιέχουν και ένα σύστημα συγκέντρωσης μιλίων κτλ. Πολύ συχνά η χρησιμοποίηση των, μάλλον ορισμένοι πιο φτωχοί, λιγότερο ευκατάστατοι καταναλωτές χρηματοδοτούν τη χρησιμοποίηση αυτών των καρτών. Προβλέπετε ότι οι έμποροι μπορούν να μην επιτρέψουν την χρησιμοποίηση των καρτών αυτών ή να θέσουν μια υψηλότερη προμήθεια για τη χρησιμοποίηση των καρτών αυτών. Τώρα, όσον αφορά το co-branding, Καταλαβαίνω ότι είπε η κυρία Εντβέλτ ότι σε κάθε περίπτωση θα δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Και ακριβώς αυτό βλέπουμε και προκειμένου. Ο βασικός κανόνας που ισχύει εδώ πέρα, οποιαδήποτε αλλαγή και να γίνει, θα πρέπει να προβλέπει το εξής ότι η οικονομία θα λειτουργεί αποτελεσματικά αν τελικά ο παράγοντας εκείνος ο οποίος πρέπει να πληρώσει για ένα προϊόν ή για μια υπηρεσία είναι και αυτός ο οποίος τελικά κάνει την τελική επιλογή, δηλαδή είτε ο καταναλωτής εν προκειμένου είτε ο έμπορος, γιατί αυτοί καταβάλουν τελικά με τον έναν άλλο τρόπο την προμήθεια. Δεν θα πρέπει μέσω του καονισμού αυτού να ευνοούνται οι τράπεζες οι οποίοι αυξάνουν τα κέρδη τους μέσω των κρυφών αυτών τελών. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέγει το μέσο το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει και ο έμπορος επίσης. Πρώτα, πρώτα ο έμπορος και έπειτα ο καταναλωτής. Και βέβαια ο καταναλωτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορεί να επιλέγει το μέσο το οποίο θέλει, να μην προαποφασίζει για αυτόν ο έμπορο. Ο πρόεδρο διακόπτη. Πρέπει να ολοκληρώσετε γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Λοιπόν, ε, ολοκληρώνω, συμφωνώ μαζί σας, ολοκληρώνω. Τελευταίο σημείο όσον αφορά τους κανόνες μη, πα, μη παράκαμψης ε, του κανονισμού αυτού. Βλέπουμε ένα αντίστοιχο κανόνα και στην Αμερικανική νομοθεσία. Ουσιαστικά θέλουμε εδώ πέρα να αποφύγουμε οι τράπεζες ή άλλα συστήματα να δημιουργήσουν μηχανισμούς που τελικά θα παρακάμψουν τις διατάξεις που προβλέπει αυτός ο κανονισμός. Ιδίως στα σημεία εκείνα που θέλουμε να αποφύγουμε, να καταργήσουμε τους κανόνες αυτούς για τις εγχώριες ή τις διασυνοριακές συναλλαγές. Εσείς θέλετε να κρατήσετε τους κανόνες αυτούς για τις εγχώριες αγορές, να τις καταργήσετε για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέμε ότι οι κανόνες αυτοί μη παράκαμψης, δηλαδή τις νομοθεσίες θα πρέπει να ισχύουν και για τις εγχώριες και για τις διεθνείς συναλλαγές. Yeah. Ευχαριστώ εσείς τώρα, για το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ναι, ναι, παρακαλώ να είσαστε σύντομο, λέει ο πρόεδρο. Δύο πράγματα θα γίνουν με την οδηγία αυτή. Θα ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή όσον αφορά τι πληρωμέ, διευρύνοντα το ευρώ εφαρμογή τη οδηγία σε οικονομικού παράγοντε, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά πληρωμών. Αλλά μέχρι τώρα ήταν αυτό μόνο με εξαιρέσει. Η μία περίπτωση είναι και οι online πληρωμές που προτείνουμε να συμπεριληφθούν και αυτές την οδηγία για τις υπηρεσίες και τις πληρωμές. Εδώ θα πρέπει να βασιστούμε βέβαια στους βατικούς όρους των πλατφόρμων αυτών. Με τέτοιο πνεύμα η πρόταση περιορίζει τις εξαιρέσεις που έχουν οι Telecom για τις πληρωμές για τους ίδιους λόγους. Η οδηγία αυτή θα ενισχύσει επίση την ασφάλεια πληρωμών, συμπεριλαμβάνοντα και τι online πληρωμέ, γιατί θα ζητάει ταυτοποίηση από πλευρά του καταναλωτή. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τι απάτε και γι' αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε το λόγο για τον οποίο το 40% των ε, πολιτών που χρησιμοποιούν ε, το διαδίκτυο δεν κάνουν αγορές online. Θέλουμε δηλαδή ένα νομικό πλαίσιο για τους ε, φορείς πληρωμών. Θέλουμε να νομοποιηθούν οι εταιρείε που λειτουργούν στην αγορά αυτή προστατεύοντας τους καταναλωτές και τους ε, λιανοπολιτές. Θα υπάρξει ένα μητρό με αυτούς που χρησιμοποιούν ε, που δέχονται τέτοιες πληρωμές. Θέλουμε καλή ισορροπία για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και των λιανοπολιτών και των καταναλωτών αλλά να λάβουμε υπόψη μας και όλες τις ε, παραμέτρους της ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Τα συστήματα πληρωμόνο πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια και αυτός είναι ο κύριος στόχος της πρότασής μας. Φυσικά μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Θέλουμε ιδιαίτερα τους ε, νέους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις πληρωμές αυτές να τους προστατεύσουμε. Για το θέμα των τελών, η πρόταση αυτή θα είναι σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις ορίων που δεν υπάρχουν ανώτατα όρια. Πάντως Ελπίζουμε ότι οι δύο συγητές ε, και πιστεύουμε θα καταλήξουν σε μια ισορροπημένη λύση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Σύντομα τώρα κάποια σχόλια έχω να κάνω και εγώ όσον αφορά την συζήτησή μας μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλιά τους. Συμφωνώ κύριε Μπαλντίνη. Πρέπει να δημιουργήσουμε πράγματι ένα ενιαίο και αποτελεσματικό σύστημα. Νομίζω ότι είναι κοινό στόχος αυτός. Και αυτά που είπε Σόφη Συμφωνώ για το ότι είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία να μην ισχύει μόνο για τα σημερινά συστήματα πληρωμών, αλλά και για τα επόμενα, τα μελλοντικά συστήματα πληρωμών. Όποια και αν είναι αυτά που εμφανιστούν αργότερα. Για το τριμερές σύστημα είμαι διατεθειμένος να συζητήσω τη δυνατότητα να βρούμε μια διατύπωση όπου θα συμπεριλάβουμε και αυτά εφόσον φτάσουν σε κάποιο επίπεδο συμμετοχή στην αγορά. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να το συζητήσουμε για να βρούμε μια λύση. Για το co-badging. Το είπε και η Σόφη και η Πράσινη και ο Σάμπο. Είναι σημαντικό σε σχέση με το πλαστικό χρήμα να βρούμε μια λύση σε προαιρετική βάση, όχι υποχρεωτική. Όσον αφορά τα άλλα συστήματα πληρωμών, νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Για το co-badging πάντως θέλω μία διατύπωση πιο συγκεκριμένη. Για τα άλλα θέματα επίσης πρέπει να βρεθεί η σωστή διατύπωση όσον αφορά το Honor All Card. Νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το μεσόρο για τις τιμές, τις απόλυτες τιμές, αντί για τις ανώτατες. Να ψάξουμε να βρούμε και εδώ μια διατύπωση που να ικανοποιεί όλους μας. Τέλος, συμφωνώ με το Σάμπο για το ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους καταναλωτές στην καθημερινή του ζωή, ώστε η ρύθμιση αυτή να τους διευκολύνει τις πληρωμές με κάρτα και όχι να πετύχουμε τον αντίθετο στόχο, δηλαδή να δυσκολέψουμε τη χρήση των καρτών αυτών πληρωμών. Επιμένω και πάλι με τις ευχαριστίες μου και προς τον συνεισηγητή μας εδώ πέρα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως με καλή βούληση θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα όσα μας προβληματίζουν σήμερα. Αποτελεσματικές και λύσεις με ισορροπημένη προσέγγιση. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Φέιο για να απαντήσει στα σχόλια που έγιναν στη δικιά του έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ και θα είμαι πολύ σύντομο στο μέτρο <clears throat> για το ότι πρέπει να πούμε ότι εδώ και μια ώρα ασχολούμαστε με αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες και τις, ε, τους θαλάμους διερμηνίας, τους διερμηνείς επίσης και να πω ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η πρόταση <clears throat> για το πιστή που παρουσιάζεται εδώ ανταποκρίνεται σε ένα σημείο αφετηρίας. Είναι μια αφετηρία. Αφετηρία η κίνηση που μου δίνει όμως και ικανοποίηση σε σχέση με τη συζήτηση που διαμορφώθηκε εδώ, σε σχέση με τις διαφορές, διαφορές μεταξύ των αγορών που πρέπει να παρατηρήσουμε και στο μέτρο του δυνατού του εφικτού να εναρμονίσουμε. Και όσον αφορά τις ε, αναφορές για τη σπουδαιότητα πληροφόρησης που θα είναι σαφής η πληροφόρηση. Υπάρχει ανάγκη να προσαρμοστούμε σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για το μέλλον, για τους νεοεισερχόμενους στις αγορές και να είναι, προσπαθήσουμε, είναι προφανές, να προβλέψουμε και να έχουμε δυνατότητα να προσαρμοστούμε και να αντιδράσουμε για τα όσα θα συμβούν στο μέλλον. Και επίσης θέλω να επιστήσω την προσοχή ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, των μέσων πληρωμών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται. Και σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση θέσεων είναι το θέμα του surcharges τη σύσπραξης των τελών. Είμαι απόλυτα ανοιχτός για τις προτάσεις και τις, ε, ε, τα σχόλιά σας οδηγηθούμε σε μια πρόταση που να ρυθμίζει αυτό το θέμα. Είμαι πρόθυμος να συζητήσω με τους συναδέλφους, με τους γιώδεις συζητητές για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια σύμφωνη θέση, τελική συμφωνία. Να πω επίσης ότι υπήρξε μία αναφορά των συναδέφων για την διορία, για την προθεσμία, για την κατάθεση τροπολογιών που βρίσκεται πολύ ε, σύντομα σε σχέση με τις ε, ε, διακοπές των Χριστουγέννων και θα πρέπει σίγουρα να συζητήσουμε με τις υπηρεσίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για να δούμε την δυνατότητα να υπάρξει μια προσαρμογή, μια τροποποίηση αυτής της προθεσμίας ίσως. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι προγραμματίζουμε ένα στρογγυλό τραπέζι στις 7 Ιανουαρίου για αυτό το θέμα. Είναι μια άλλη ευκαιρία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ιδέες μας για αυτό το θέμα. Και το βρίσκω θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρουσίαση που έγινε ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι η ώρα το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν να κάνει αυτό το οποίο είναι αναγκαίο και να συνομιλήσει με τα θεσμικά όργανα το Ευρωκοινοβούλιο ώστε να υπάρξει αυτή η ε, αφετηρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί. Θα συναντηθούμε στι 3. Α, η προθεσμία θα είναι 9 Ιανουαρίου. Η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στις 12 ή 13 Φεβρουαρίου του 2014 και θα ψηφίσουμε προσέγγιση στην Επιτροπή Οικονομίας ε, ε, Οικονομικών στις 20 Φεβρουαρίου και θα περάσουμε στην Ολομέλεια στην περίοδο συνόδου του Απριλίου. Μα, ίσως έτσι θα καταφέρουμε. Και ολοκληρώνουμε εδώ τις εργασίες μας μέχρι τις 3 το απόγευμα στην ίδια αυτή αίθουσα. Ευχαριστώ όλους σας. Γεια σας.